σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Συνεχίζουμε την συνεδρίαση. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας για τα BEPP, τα Πανευρωπαϊκά Ευρωπαϊκά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προσπαθήσει να θέσει σε συζήτηση το θέμα του Ευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού προϊόντος ήδη από το, 2016. Σήμερα θα ασχοληθούμε για τις πρακτικές επιπτώσεις των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τίνουν να δημιουργήσουν ένα νέο ευρωπαϊκό μέσο. Αυτό αναφέρεται και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 για την χρηματοδότηση των συντάξεων και για την ενίσχυση των κεφαλαίων έτσι ώστε να υπάρξει στροφή περισσότερων ε, από μεγαλύτερης αποταμίευσης προς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και θα πρέπει χρησιμοποιώντας τα κοινά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις συνθήκες που ισχύουν σε κάθε χώρα να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό ενός ενιαίου τέτοιου είδους προϊόντος. Η πρόταση συνοδεύεται από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογική αντιμετώπιση του προϊόντος αυτό. Ενθαρρύνονται τα κράτη-μέλη να ε, καθιερώσουν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και αυτό είναι προϋπόθεση της επιτυχίας του συνταξιοδοτικού αυτού του μέσου. Θα ακούσουμε κάποιους ε, εκπροσώπους ασφαλιστικών εταιριών, πανεπιστημίων, συνταξιοδοτικών ταμείων και οργανώσεων των πολιτών. Κάθε ομιλητής παρακαλώ για πέντε λεπτά. Ε, αμέσως μετά θα υπάρξουν ερωτήσεις από τα μέλη δύο λεπτά το κάθε ε, μέλος ε, για να θέσει το ερώτημά του. Δεν θέλω άλλο από το χρόνο σας. Ο πρώτος ομιλητής για σήμερα είναι ο κύριος Τόμπιας Μπίχλερ από την ασφαλιστική εταιρεία Allianz Γερμανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρουσιάσω την θέση μας για το Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν. Η Allianz πρέπει να πω γενικά στηρίζει την ε, εισαγωγή ενός τέτοιου πανευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού προϊόντος <clears throat> στα πλαίσια ενός καλά σχεδιασμένου δεύτερου καθεστώτος για να αναπτυχθεί η Ένωση Κεφαλαία Αγορών Πιστεύουμε ότι έτσι θα κλείσει το συνταξιοδοτικό κενό που υπάρχει στην Ευρώπη, θα προωθηθεί η ανάπτυξη με επενδύσεις στην πραγματική οικονομία στην Ευρώπη που θα είναι και μακροχρόνιες. Γι' αυτό η Αλιάνσε εργάστηκε επικοδομητικά με σημαντικούς εμπλεκομένους τους προηγούμενους μήνες και με τη δική μας εταιρεία και με ιδιωτικές εταιρείες και με δημόσιες. Συζητούμε τις δικές μας απόψεις για το πανευρωπαϊκό προϊόν με όλες τις εταιρείες όπου υπάρχουν, εμείς έχουμε υποκαταστήματα σχεδόν παντού, έχουμε και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και έχουμε ένα, ε, μια πλήρη, μπορώ να πω, εποπτεία της αγοράς εν προκειμένου. Για την τωρινή πρόταση, Βλέπουμε σημαντικές προκλήσεις στην ε, πρόταση. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι δεν είναι η πρόταση αυτή πανευρωπαϊκή, ούτε παρέχει συνταξιοδοτικό προϊόν. Να συγκεκριμενοποιήσω. Δεν είναι συνταξιοδοτικό προϊόν γιατί η φάση αποσυσσόρευσης σύνταξης δεν καλύπτεται αρκετά στην πρόταση ως έχει. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα μιλάμε για ένα αποταμιευτικό προϊόν, αν περί αυτού πρόκειται τότε πρέπει να του βρούμε και άλλο όνομα αλλά από, εμείς πιστεύουμε ότι η φάση αποσυσσόρευσης σύνταξης θα πρέπει να ρυθμίζεται πάρα πολύ προσεκτικά από τον κανονισμό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερον, δεν είναι πανευρωπαϊκή. Αυτό θα σας εκπλήξει που το λέμε, αλλά αυτό έχει να κάνει με την πρόταση που είδαμε και που αφορά επιμέρους τομείς ή τμήματα στο ΠΕΠ. Η τωρινή πρόταση ουσιαστικά ε, ζητεί από όλους τους παρόχους να παρέχουν σε κάθε κράτος μέλος συγκεκριμένο τομέα που αντικατοπτρίζει τις τοπικές συνθήκες σε επίπεδο κυρίως φορολογικό στα κράτη-μέλη. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό σε τελευταία ανάλυση θα οδηγήσει στο εξής. Θα έχουμε συνδυασμό υφισταμένων τοπικών προϊόντων αντί για το λεγόμενο πανευρωπαϊκό σου generis προϊόν. Και εμείς αυτό θέλαμε να είχε γίνει. Αυτό θεωρήσαμε ότι σε αυτό απέβλεπε το ΠΕΠ. Αυτά λοιπόν είναι δύο σημαντικά θέματα που πρέπει να λυθούν τους επόμενους μήνες. ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η πρόταση, για να το πω έτσι. Τώρα, αν μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ και λαμβάνοντας υπόψη την ε, δημιουργία αξίας ε, για τους ε, πελάτες και υγιή ανταγωνισμό, πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία που ο κανονισμός ΠΕΠ πρέπει να ρυθμίσει εις ό,τι αφορά τα ελάχιστα πρότυπα σε πανευρωπαϊκή βάση. Η τωρινή πρόταση αφήνει πολύ διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη. Εμείς θα θέλαμε ένα δεύτερο ή δευτερογενές καθεστώς, το οποίο θα ορίζει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Ε, για να μην μακρηγορήσω, ε, για τις εγγυήσεις πιστεύουμε ότι ε, η ε, τα ταμεία εγγυήσεων ε, έχουν μια ε, εγγύηση κεφαλαίων, αλλά δεν διευκρινίζεται τι σημαίνει αυτό ιδιαίτερα σε φάση διατομεακή. Η εγγύηση ασφαλιστική εταιρεία διαφέρει από προϊόντα ενός κύκλου ζωής που θα αντιμετωπίζονται από διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και εκεί είναι δύσκολες οι εγγύησεις. Βέβαια, εδώ μιλάμε για ίσως, ισότιμους κανόνες ανταγωνισμού. Οπότε αυτό δεν ε, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου. Για τις εγγύσεις θα πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς κατάλληλο. Εμείς το επεξεργαζόμεθα εδώ και χρόνια και έχουμε καταλήξει το 2016 κάπου. Θα το συζητήσουμε αυτό. Επίσης, να μιλήσω και για την προστασία του καταναλωτή, του πελάτη ε, και τη διαφάνεια. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις ήδη εδώ για το πώς δίνουμε πληροφορίες και πώς προστατεύουμε τους πελάτες μας. Ε, αν ε, το ΠΕΠ θα έχει κάποιες βασικές εγγυήσεις, αλλά προσφέρεται στα κράτη-μέλη και από τις διάφορες εταιρείες με διαφορετικές προϋποθέσεις, αυτό πρέπει να το δούμε. Για την αποσυσσόρευση μίλησα, ε, στην αρχή τουλάχιστον 50% ε, των αποταμιεύσεων θα πρέπει να επενδύονται σε ένα προϊόν που θα έχει αιτήσει απόδοση και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό δεδομένου ότι ε, αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής στην Ευρώπη. Ε, γιατί ε, το 80 με 90% ε, ε, των δυνητικών υποψηφίων για ένα τέτοιο προϊόν θα εμείωναν αν ρωτώνται το προσδόκιμο ζωής. Επίσης, για την αλλαγή ε, μεταξύ από πάροχο σε πάροχο ή από προϊόν σε προϊόν ε, χρειάζονται ενιαίοι κανόνες και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το περιορίσουμε στην τωρινή αγοραία αξία του προϊόντος μέχρι τη συνταξιοδότηση. Δηλαδή, ε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην δημιουργήσουμε αντικίνητρα στο προϊόν αυτό και να ε, υπάρξουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Δηλαδή να μην ε, υπάρχουν αποχωρήσεις μετά από ας πούμε μία πενταετία. Τέλος, σημαντικό αυτό, εμείς ε, γενικά στηρίζουμε την ιδέα του πανευρωπαϊκού συνταξιδοτικού προϊόντος. Ανέφερα βέβαια κάποιες δυσκολίες που βλέπουμε, αλλά επίσης και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται εδώ, και το έχω πει αυτό σε διμερείς συναντήσεις, και αυτό είναι δύσκολο, για να το πω ήπια, όταν μιλάμε για το Solvency 2 και ε, ε, εδώ μιλάμε για ένα διατομεακό προϊόν, το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζει εκατομμύρια ε, ενδιαφερομένους. Με αυτές τις παρατηρήσεις κλείνω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να τηρείτε παρακαλώ το χρόνο για να προλάβουν όλοι οι ομιλητές, γιατί μετά θα πρέπει να ε, λάβουν το λόγο και ο εισηγητής και η σκιώδης. Ε, ο δεύτερος ε, ομιλητής μας είναι ο Μπερνάρα Γκυγιόν ε, από την Αμούντι, επικεφαλής των διακανονισμών. Ε, ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθώ στο θέμα αυτό, με το οποίο το Αμούντι ασχολείται εδώ και πολύ καιρό. Ασχολούμεθα με τα θέματα συμπληρωματικότητας των συνταξιοδοτικών προϊόντων και γι' αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ΠΕΠ. Το ΠΕΠ έχει τρεις βασικούς στόχους θα έλεγα. Το πρώτο είναι να εμπλουτιστεί η προσφορά ε, δημόσιων και επαγγελματικών συντάξεων με νέα προϊόντα υψηλής αξίας έτσι ώστε να βελτιωθεί η, η βιωσιμότητα, αν θέλετε, η οικονομική των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Ταυτόχρονα να στραφούν κάποιες μορφές αποταμίωσης σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα, αυτός άλλωστε είναι ένας βασικός στόχος της Ένωσης Κεφαλαίων. Να προσθέσω επίσης ότι η προετοιμασία της συνταξιοδότησης είναι το αντικείμενο της ε, αποταμίευσης. Και ο τρίτος στόχος, ίσως ο πιο σημαντικός, είναι να υπάρξει μια λύση συνταξιοδοτική για τους κινητικούς πολίτες. Αυτό ακριβώς καλύπτεται και από το επίθετο πανευρωπαϊκός. Σχετικά με τον πρώτο στόχο τώρα, η κατάσταση των επιτοκίων στην Ευρώπη και η μακρά διάρκεια ζωής των Ευρωπαίων πολιτών μας υποχρεώνει να αποκλίνουμε από τα παραδοσιακά ασφαλιστικά σχήματα. Αυτά τουλάχιστον στην Γαλλία στην οποία αναφέρομαι κυριαρχείται από επενδύσεις στον τομέα των ομολόγων. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί οποιαδήποτε λύση η οποία θα αναζητήσει να επιβάλλει μια επίσημη εγγύηση θα οδηγήσει στην υποχρέωση ε, ε, επένδυσης σε ομολογίες έτσι ώστε να μειωθεί ε, το κόστος αυτών των εγγύσεων. Η εναλλακτική πρόταση σε σχέση με τις σταδιακές αυτές απομακρύνσεις σταδιακές από τον κίνδυνο είναι κάτι το οποίο θα συνδυάζει και τους στόχους προστασίας από τις εξωτερικές αρνητικές συγκυρίες όπως επίσης και από τις υπεραποδόσεις σε ορισμένες χρονικές φάσεις. Ε, νομίζω ότι τα τεστ τα οποία έχουμε κάνει στο Αμούντι δείχνουν ότι οι πιθανότητες να συναντηθούν τέτοιες περίοδοι στη ζωή ενός επενδυτικού προϊόντος είναι πάνω από 90%. Μία πανεπιστημιακή μελέτη γύρω από το θέμα αυτό σύντομα θα μας δώσει στοιχεία και θα δοθεί και στην εφάμα Στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, οι ε, μελέτες αυτές ε, υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια και δίνουν νομίζω πολύ ενημερωτικά αποτελέσματα. Ο δεύτερος στόχος είναι οι μακροπρόθεσμες μορφές αποταμίευσης. Μακροπρόθεσμες επενδύσεις οι οποίες χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία όπως επίσης και ε, υψηλά ασφάλιστρα για τους, και αποδόσεις για τους επενδυτές. Ε, μετοχές αλλά ταυτόχρονα και ε, υποδομές ή επίσης και επενδύσεις στον τομέα των κατοικιών και των, της οικοδομής γενικότερα και βασικός τελικά ο στόχος είναι να υπάρξει λύση και για τους ε, ε, κινητικούς εργαζομένους που θα μπορούν να μεταφέρουν το προϊόν τους από τη μία χώρα στην άλλη. Το, η ύπαρξη και η χρήση των τμήματων, των επιμέρους τμήματων στην διαδικασία σώρευσης της σύνταξης είναι μια λύση για την αμόντι. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με απλό τρόπο για τους επενδυτές αλλά όχι πάρα πολύ απλό για τους παρόχους. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την υποχρέωση για όλους τους παρόχους να έχουν 27 διαφορετικά κομπάρτμαν σε κάθε περίπτωση ασφαλιστικού συμβουλίου. Η Αμούντι είναι παγκόσμιος παίκτη. όλα αυτά έχουμε 7 ή 8 τμήματα για κάθε ένα από τα συνταξιοδοτικά προγράμματα σύμφωνα με την οδηγία της Επιτροπής. Είναι λοιπόν αδύνατο για τους μικρούς παρόχους να δημιουργήσουν αυτά τα 27 τμήματα και δεν θα είχε και πραγματικό νόημα. Συν της άλλης θα στερήσει από μικρές χώρες την ύπαρξη τοπικών παρόχων ενιαίων ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία σε σχέση με την πρόταση αυτή και να λάβουμε υπόψη μας τις ισορροπίες και ανάμεσα στις χώρες που ανήκουν στην ίδια ευρύτερη περιφέρεια. Σας ευχαριστώ. Καθηγητής Φαν Μίρτεν από την Ουτρέχτη, το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Ευχαριστώ. Η παρουσίαση μου αφορά την δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιωτικών ε, σχημάτων με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο που είναι και η ειδικότητά μου σημειώνω ότι πολλές συζητήσεις στηρίζονται σε εσφαλμένες παραδοχές τρεις συγκεκριμένα πρώτον ότι η ΟΡΠ δεν είναι οικονομικές ε, επιχειρήσεις δεύτερον ότι είναι αντίθετο ένα τέτοιο σχέδιο με δευτερεογενείς δραστηριότητες και τρίτον ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχήμα χωρίς αρμονισμένο φορολογικό σύστημα. Είναι σφαλμένες λοιπόν και οι τρεις ε, παραδοχές και θα εξηγήσω γιατί. Δεν είναι λοιπόν χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις λένε οι ORPS και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες. Αυτό είναι ασφαλμένο διότι παραδείγματι η γερμανική BPI είναι μια τέτοια επιχείρηση δεύτερο πυλώνα πλήρως αναπτυγμένη χρηματοοικονομική χρηματοπιστωτική επιχείρηση. Γιατί να αποκλειστούν λοιπόν. Ξέρω ότι είναι πολύ έντονο το λόμπι που γίνεται αυτή τη στιγμή για να αποκλειστούν οι ΙΟΡΠΣ e από το ΠΕΠ. E Πράγμα το οποίο θα ήταν ασφαλμένο. Ξέρετε ότι η οδηγία η e 2 κάνει μια διάκριση που προβλέπει την δραστηριοποίηση Φερρυπίν στην ε, Ολλανδική αγορά, δηλαδή επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση και άρα δεν μπορούν να αποκλειστούν ε, εκ προημίου ή ΟΡΠ. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε στον αποκλεισμό των ΙΟΡΠ και νομίζω τρία χρόνια πριν είχε γίνει μια ε, ακρόαση για την ΙΟΡΠ 2 στην οποία επίσης είχα λάβει το λόγο, αναπτύσσοντας την ιδέα ότι μπορεί να αποκλειστούν μόνο αυτές οι όρπ οι οποίες δεν είναι κοινέ, ε, δεν καλύπτονται από το ΙΟΡΠ e αφενός και δεν ε, δραστηριοποιούνται πέραν των συνόρων. Αυτό δεν το προέβλεψε δυστυχώς η οδηγία, αλλά ίσως θα ήταν αυτό μια ιδέα. Να αποκλειστούν μόνο οι ΙΟΡΠ e που δεν έχουν διασυνοριακές δραστηριότητες και δεν έχουν χρηματοπιστωτικό χαρακτήρα. Γιατί μπορεί να γίνει αυτή η διαφοροποίηση. Μπορείτε να δείτε τις τροπολογίες του κύριου Τάνι, παραδείγματι, για την οδηγία ΙΟΡΠ. Δεύτερο επιχείρημα ότι το ΠΕΠ ε, είναι αντίθετο με τις δευτερογενείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Από πλευράς του ευρωπαϊκού δικαίου, το ΠΕΠ δεν είναι δεύτερο πυλόν, επομένω δεν μπορεί να είναι αντίθετο με τις δευτερογενείς δραστηριότητες. Η οδηγία 2 στο άρθρο 7 λέει ότι τα τα ταμεία που προσφέρουν ε, πλεονεκτήματα κέρδος και δραστηριότητες ε, δεν θα πρέπει να αποκλειστούν. Επομένως το ΠΕΠ εδώ εντάσσεται ωραιότατα στις δραστηριότητες του ΝΙΟΡΠ. Η τρίτη παραδοχή που ακούγεται είναι ότι το ΠΕΠ δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ένα αρμονισμένο φορολογικό σύστημα. Δύο λόγια εδώ. Καταρχάς είναι η πρώτη φορά στον κανονισμό ΠΕΠ που κάλυψε το θέμα της δυνατότητας μεταφοράς για πρώτη φορά σε ατομικό και σε συλλογική βάση, δηλαδή στην ΙΟΡΠ 2 βλέπουμε συλλογικές μεταφορές δικαιωμάτων που καθιστούν ακόμη και πιο δύσκολο θα έλεγα, όχι πιο εύκολο να μεταφερθούν τα ποσά. Και έτσι έρχομαι στο θεμελιώδες ερώτημα. Τεθνικά νομοθετήματα είναι αντίθετα στην ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όντω. Πρέπει ένας ε, πολίτης να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα συνταξιωτικά του δικαιώματα μαζί. Εάν οι εθνικές όμως δετάξεις de facto το αποκλείουν αυτό, Μήπως είναι και οι φορολογικές διατάξεις αντίθετες με την ελεύθερη διακίνηση. Στον κανονισμό ΠΕΡΠ νομίζω μπορούμε να έχουμε την ε, ελαχιστοποίηση των συνεπειών των διαφορετικών φορολογικών συστημάτων. Δηλαδή δυνατότητα μεταφοράς χωρίς πραγματική δυνατότητα μεταφοράς. Μπορεί κανείς να τοποθετήσει ποσά στο πρώτο τμήμα, compartment 1, χωρίς μεταφορά του στο compartment 2, που υπάγεται στο δίκαιο άλλου κράτου μέλου. Αν κάποιο στην ηλικία των 67 παραδείγματα έχει ταξιδοτηθεί, θα πρέπει να μπορεί να συνενώνει τα διαφορετικά compartments. Άρα δεν χρειάζεται να φορολογηθούν διαφορετικά τα διαφορετικά compartments. Επίσης λέγεται ότι διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα εφαρμόζονται σε διαφορετικά compartments, αλλά και στις κατοχώρες έχουμε συστήματα BP, SD, τα λοιπά Και δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο επικυρώνεται το επιχείρημα ότι χρειάζεται μια φορολογική αντιμετώπιση. Επίσης, και με κάθε σεβασμό σε όσους έχουν κάνει τις προσπάθειες, ε, στο θέμα αυτό η ΕΟΡΠ δεν επιτρέπει πραγματική δυνατότητα μετακίνησης και άρα ε, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο ΕΟΡΠ, στο ΠΕΡΠ. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η Άννα Φίλη, η οποία εκπροσωπεί τις Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Καταναλωτών BUC. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΟΝ που εκάλεσε την BUC να συμμετάσχει. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές όλο και περισσότερο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνταξιδοτικές τους ανάγκες στα πλαίσια της αποδυναμωνόμενης οικονομίας, δημοσιονομικών περιορισμών, ε, επιδιώκουν προσωπικά προϊόντα. Είναι αρκετά ε, περίπλοκη η κατάσταση, όπως και το κόστος των προϊόντων. Ε, είναι ε, πολύ ε, σημαντικό λοιπόν να χαιρετήσουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν επιτύχει. Το ΠΕΠ θα βοηθήσει να μειωθούν κάποιες ανεπάρκειες στην αγορά. Θα δημιουργηθούν τυποποιημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα και θα βελτιωθεί η ε, αγορά των επενδύσεων ε, λιανικής. Ε, έτσι, τα, τη, βέβαια, πολλές φορές τα προϊόντα που υπάρχουν ήδη μπορούν να καλυφθούν από νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος. Ε, υπάρχουν κάποια θέματα που θα ήθελα να αναφέρω. Καταρχήν η επιλογή εγγυημένων επενδύσεων. Πιστεύουμε ότι είναι ε, σημαντικό αυτό το χαρακτηριστικό του ΠΕΠ, ε, υποχρεωτική ε, πρόβλεψη για μια τέτοια επιλογή. Αυτό έχει μεγάλες δυνατότητες για καταναλωτές που δεν μπορούν να κάνουν μια ενημερωμένη επιλογή όταν αποταμιεύουν για την συνταξιοδότηση. Ε, είναι πολύ σημαντικό επίσης να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ε, ε, ανθρώπων που έχουν να κατανοήσουν σύνθετες πληροφορίες. Μια πιο παρεμβατική προσέγγιση είναι σημαντική για να υπάρχει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η BUC δεν είναι υπέρ των υποχρεωτικών εγγυήσεων. Το άρθρο 37 αναφέρεται στην κεφαλαιακή προστασία. Δεν είναι σαφές τι εννοεί το κεφάλαιο που έχει, που έχει επενδυθεί στο ΠΕΠ ή το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί αφού αφαιρεθούν οι διάφορες επιβαρύνσεις που χρεώνονται για το ΠΕΠ. Ε, αν το κεφάλαιο ε, είναι ε, μετά τις επιβαρύνσεις, αυτό είναι λίγο παραπλανητικό, αν εννοείται αυτό, γιατί μόνο 70% των αποταμιεύσεων που έχουν συσσωρευτεί θα προστατεύονται και μόνο ονομαστικά. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ε, τις εγγυήσεις και αν χρειάζεται να ενσωματωθούν. Ε, πολλές φορές ε, έτσι η συνθετότητα του προϊόντος ε, αυξάνεται και είναι, υπάρχουν επενδύσεις χαμηλής απόδοσης. Δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την μακρά διάρκεια των προϊόν, του προϊόντος ΠΕΠ και τις πληθωριστικές πιέσεις. Καμιά φορά μπορεί να είναι καλές οι εγγυήσει όταν ο, είναι κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης δεν είναι καλές οι παντού. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ε, υπάρχει ε, μια επιλογή για τα μία εγγύησεων και κάθε επιλογή θα πρέπει να εξηγείται σαφώς τον ε, καταναλωτή. Τώρα για το κόστος. Το ΠΕΠ και τα συναφή προϊόντα είναι τα πανηρά και σύνθετα. Ε, επίσης υπάρχουν πάρα πολλές ε, ε, χρεώσεις επιβαρύνσεις κατά τη διάρκεια του προϊόντος που επηρεάζουν την αποδοτικότητά του. Ας πούμε για ασφάλιστρο 100 ευρώ που επενδύεται σε ένα προϊόν συνταξιοδοτικό στην Αυστρία από τα 100 μόνο τα 70 ευρώ πηγαίνουν στις αποταμιεύσεις τα πρώτα 5 χρόνια και μετά το πέμπτο έτος ε, το ποσοστό του ασφαλίστρου που πηγαίνει στις αποταμιεύσεις είναι 84 ευρώ. Ε, η καθαρή απόδοση λοιπόν είναι κοντά στο 0, ακόμα και αρνητικό μπορεί να είναι λόγω των υψηλών χρεώσεων. Το υψηλό κόστος δεν αναφέρεται στην πρόταση, αλλά στο βαθμό που θα πληρώνουν ε, υψηλές χρεώσεις δεν υπάρχει κίνητρο να επιλέξουν ένα ΠΕΠ οι καταναλωτές. Γι' αυτό ε, θα πρέπει ε, να, να, υπάρξει διάταξη η οποία θα θέτει ανώτατο όριο στις χρεώσεις, στις προμήθειες και τα άλλα κόστη. Και θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες επιλογές γι' αυτό. Επίσης, η διαδικασία ε, έγκρισης, αδειοδότησης, ε, χαιρετίζουμε τον μηχανισμό που προβλέπεται, ιδιαίτερα γιατί θα είναι μία η αρχή, η ΟΠΑ, η οποία ε, θα δίνει τις άδειες. Ε, έτσι θα διευκρινίζεται το προϊόν και θα είναι ε, ανταγωνιστικό. Επίσης, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πέπ Key ID, Key Information Document. Αυτό θα πρέπει να είναι παρόμοιο με το Key ID που υπάρχει στα PRIPS και θα διευκολύνει την συγκρισιμότητα με άλλα παρόμοια ε, καθεστώτα συνταξιοδότησης ε, που υπάγονται στο PRIP Key ID. Τέλος, για την αλλαγή χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα να αλλάζουν παρόχους και προϊόντα, ιδιαίτερα ε, λόγω της μακράς διάρκειας του ΠΕΠ και της ε, ε, ανάγκης να υπάρχει πρόσβαση σε καλύτερες προσφορές στην αγορά. Ε, ε, πιστεύουμε ότι το 1,5, ε, ε, ο περιορισμός δηλαδή των συνολικών επιβαρύνσεων είναι υψηλό. Γενικά είναι καλή η πρόταση, αλλά θα πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, ο Άλουιν Ερλμανς. από μια ασφαλιστική εταιρεία με 4 εκατομμύρια πελάτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ΠΕΠ μπορεί να είναι μια χρήσιμη προσθήκη στον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα. Ο ρόλος των κρατών μελών όμως είναι κρίσιμος και θα πετύχουμε περισσότερα παραδεχόμενοι ότι ο ρόλος αυτός είναι σημαντικός. Το θέμα της συμπερίληψης ή μη των IORP ως παρόχους ΠΕΠ είναι κάτι το οποίο όχι, θα χαρακτήριζα όχι πολύ σημαντικό. Ε, νομίζω ότι εδώ έχουν περισσότερο κοινωνικό ρόλο και όχι τόσο εμπορικό θα έλεγα λόγω ύπαρξης. Ε, μεγάλοι παρόχοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν και άλλα μέσα και όχι τόσο τα IORP. Η APG σαν παράδειγμα παρέχει την δυνατότητα διαδικασίας σόρευσης ενός τέτοιου προϊόντος, ο τρίτο πυλώνα, προσφέρεται μέσα από το διαδίκτυο, το ZZPE NL είναι κάτι το ευέλικτο, το εύκολο και έχει χαμηλό ε, κόστος, 0,35 ε, κόστος ε, διαχείρισης, 35 ευρώ δηλαδή σε αιτήσια βάση και θα επανέλθω σε αυτό. Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να υποκύψει στην πρόκληση να επιβαρύνει το προϊόν αυτό με διάφορα εξωτερικά στοιχεία και θα πρέπει οι οδηγίες να δίδονται αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τις μακροπρόθεσμες ιδιαίτερα επενδύσεις στον τομέα των τραπεζών. Ε, και νομίζω ότι οι αποδόσεις έτσι και αλλιώς είναι χαμηλές λόγω των χαμηλών επιτοκίων σήμερα. Το να ζητήσει κανείς από τα ΠΕΠ να χειρίζονται τα νομικά καθεστώτα όλων των κρατών μελών μετά από τρία χρόνια λειτουργίας είναι κάτι που δεν είναι απαραίτητο, έχει πολύ υψηλό κόστος και θα εμποδίσει πάρα πολλούς παρόχους να μπουν στην αγορά. Γι' αυτό λοιπόν στοχεύουν τα ΠΕΠ να καλύψουν τις ανάγκες των τρίτο πυλώνα και μόνο θα έλεγα ο φορολογικός νόμος θα πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη. Και όλα θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον τοπικό φυσικά φορολογικό νόμο της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται το συγκεκριμένο ταμείο. Η πραγματική πρόκληση για την επιτυχία των ΠΕΠ είναι τα ακίνητρα για τα φορολογικά, επίσης η προσέλκυση νέων πελατών και αυτό θα οδηγήσει στο να δημιουργηθεί μια υγιής θα έλεγα αγορά. Εμείς έχουμε προτείνει προϊόντα που καλύπτουν περίπου το 10% των αυτοαπασχολούμενων στην Ολλανδία, 10% του εργασιακού δυναμικού. Είμαστε ο μεγαλύτερος παροχέας ενός τέτοιου προϊόντος. Θα ήθελα να πω ότι οι αυτοαπασχολούμενοι δεν είναι άνθρωποι που θα μπορέσει εύκολα κανείς να τους προσελκύσει. Θα εξοικονομούν και θα επενδύουν αλλά στα πλαίσια της περιμέτρου των φορολογικών κινήτρων. Απαιτείται περισσότερος χρόνος λοιπόν για την ανάπτυξη αυτής της αγοράς. Λύσεις fintech μπορεί επίσης να ανοίξουν νέες δυνατότητες. Όπως δείχνει η εμπειρία της APG, τα κίνητρα, τα φορολογικά είναι κάτι το σημαντικό. Δεν θα βοηθήσουν μόνο τους παρόχους να, να προχωρήσουν στην αναζήτηση των κατάλληλων φορολογικών κινήτρων σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να δηλώνουν προς την ΑΙΟΠΑ την δραστηριοποίησή τους και οι πληροφορίες αυτές νομίζω ότι θα είναι χρήσιμες για όλους. Τα κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να ωφεληθούν από τις πρωτοβουλίες ΠΕΠ θα πρέπει να οδηγήσουν τους πολίτες να συμμετέχουν σε προϊόντα όπως τα ΠΕΠ. Νομίζω ότι αυτό βλέπουμε στα πλαίσια του τι συμβαίνει στον δεύτερο πυλώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο με το λεγόμενο NEST και την λεγόμενη αυτόματη εγγραφή ή αυτόματη συμμετοχή. Και η φιλοδοξία είναι να δημιουργηθεί ένα καλύτερο εσωτερικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Η ιδέα είναι ότι αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να νομοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα εθνικά ε, συνταξιοδοτικά συστήματα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, η Επιτροπή μπορεί να κάνει βέβαια κάποιες συστάσεις να ληφθεί υπόψη στο ευρωπαϊκό εξάμεινο η σύσταση αυτή ή να υπάρξει μια αιτιολογική σκέψη στα πλαίσια ε, της απόφασης για το ΠΕΠ. Εμείς θα συνεχίσουμε να συμμεριζόμεθα την εμπειρία μας με το Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στους σκιώδεις και τους συζητητές. Μέχρι δύο λεπτά παρακαλώ ο καθένας για τις ερωτήσεις για να έχουν από τρία λεπτά οι δικοί μας να απαντήσουν. Η κυρία Αντφέλτ, Άλντε. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομη και θα αφήσω το μέσο δυνατό χρόνο για τη συζήτηση. Είμαι ευγνώμων στα πλούσια σχόλια και παρατηρήσεις των ομιλητών μας. Όλοι τους πιστεύω υπεγράμμισαν πόσο περίπλοκο είναι το θέμα πέραν βέβαια των πολιτικών επιλογών που πάντα υπάρχουν, αν δεν είναι κομματικές μπορεί να είναι εθνικές πολιτικές επιλογές, πέραν αυτού πάλι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Όταν είπε ο κύριος Μπιούχερερ ότι ήταν το χρονοδιάγραμμα πιεστικό, ήταν ευγενής βέβαια, βέβαια καλή και η πρόκληση, καλή και η δυσκολία. Δεν ξέρω αν θα καταλήξουμε όπως θέλουμε. Αλλά πιστεύω και η κυρία Φίλ νομίζω ήταν εκείνη η οποία είπε πως αν μπορέσουμε να βρούμε καλές λύσεις και καλές προτάσεις μπορούμε έτσι να στρώσουμε το δρόμο και για άλλα προϊόντα ή ρυθμίσεις. Προτιμώ να ακούσω τις απόψεις αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε φάση διαβουλεύσεων με πολλούς ε, παραγόντες και συντελεστές. Ε, θα συνεργαστώ βεβαίως με τους κοιόδης, τους ε, συντάκτες ομοδοτήσεων των άλλων επιτροπών και ελπίζω να συμφωνήσουμε σε ένα κείμενο έκθεσης για το Κοινοβούλιο, το οποίο θα εκριθεί με ευρύτατη πλειοψηφία και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε. Βεβαίω και έχω τι επαφέ με τα κράτη-μέλη που και από πλευρά του μελετούν την υπόθεση, αντιμετωπίζουν αντίστοιχε με εμά δυσκολίε. Θα βρούμε κάποιε λύσει για το εάν ε, θα περιλαϊφθούν τα ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίε περιβαλλοντικών και εξωτικών παροχών ή όχι, ε, τα compartments, οι εγγύσει κεφαλαίου, αδειοδότηση. Όλα αυτά αποτελούν μακροσκελή κατάλογο και βεβαίως τα κρατη έχουν το καθένα δικό του σύστημα για κάθε τομέα, για κάθε πάροχο με τις ιδιαιτερότητές του ο καθένας. Αλλά αν δεν κοιτάξουμε την ουσία των δυσκολιών δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε τη λύση. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ την Σοφίνετ Φέλτ. Δεν είδα, δεν άκουσα μάλλον ερώτηση, απλώς ε, απόψε. Ο κύριος Χέις, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλωσορίζω όλους ε, τους συγκεκριμένους μας εδώ. Είναι πολύ σημαντική η ακρόαση. Καταρχάς θα συμφωνήσω με την εισηγήτρια, είναι περίπλοκος ο τομέας και πρέπει να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη βεβαιότητα εδώ, να μην επιδεινωθεί η κατάσταση, γιατί όπως έχουμε πει ήδη με τα ΙΟΡΠ, τα Ιδρύματα Προσφέρων Υπηρεσίας Επαγγελματικών Στρατιωτικών Παραχών, ε, παίρνουμε αποφάσεις για τα χρήματα των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να γίνει ο σχεδιασμό σωστά, ώστε να μην μετατραπεί αυτό το πρόγραμμα, αυτή η λύση, σε μια λύση που κανείς δεν δέχεται να υιοθετήσει. Και βεβαίως μας απασχολεί το θέμα της προστασία των καταναλωτών και τα θεμελιώδη ζητήματα των ε, υπερβολικά ακριβών τελών, ε, επιβαρύνσεων, ε, τιμών κτλ. Από την άλλη βεβαίως θα πρέπει να προσφέρεται και μια γκάμα προϊόντος ικανοποιητική. Πρέπει να δώσουμε αρκετό χρόνο, έστω και αν είναι φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα, και πάνω απ' όλα να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να είναι σωστή η περιγραφή, ο σχεδιασμός του προϊόντος με βάση τους στόχους μας και τις απαιτήσει μας κύριος Μάρτεν ε, είπε ότι δεν θα φέρει μεγάλη διαφορά ως προς τις ε, ε, επιχειρήσεις και την εγκαθίδρυση τους υπερσυνοριακά η εορτ 2. Νομίζω ότι είναι νωρίς αυτό γιατί ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά σε εθνικό δίκαιο της οδηγίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς σε αυτό το στάδιο να κάνει τις δηλώσεις. Επίσης, το ζήτημα της πλήρους χρηματοδότησης που ήταν ε, πρόβλημα στην πρώτη ΕΟΡΠ και το ζήτημα της ε, ασφάλειας ως προς τον ε, πάροχο της χώρας προελεύσεως και υποδοχής που επίσης θα πρέπει να ρυθμιστεί. Τρία συγκεκριμένα ερωτήματα λοιπόν για την ΑΕΟΠΑ. Θα ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες όλους, εάν είναι ο κατάλληλος φορέας. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι είναι πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό σώμα για ένα πανευρωπαϊκό ε, προϊόν. Θα ήταν σκόπιμο να απευθύνεται κανείς στην ΕΟΠΑ. Αλλά από την άλλη πολλές αποφάσεις θα λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη. Μήπως, παρακαλώ κύριε συνάδελφε στο μικρόφωνο. Ναι, μήπως τελικά όμως επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το τελικό αποτέλεσμα των απευθυνόμαστε στην ΕΟΠΑ. Έχω εγώ βέβαια την άποψή μου, αλλά θέλω και τις δικές σας. Δεύτερον, εγγύηση έναντι μιας ανοιχτή επιλογής και ζωή Μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το συνδυασμό και να τον προσαρμόσουμε στις ανάγκες των καταναλωτών γιατί βέβαια θα, πάρουν, θα αναλάβουν εγγυήσει ή θα επιλέξουν εγγυήσει οι περισσότεροι πολίτε καταναλωτέ, γιατί δεν θα γνωρίζουν τι θα γίνεται μακροπρόθεσμα. Αλλά μήπω με τι εγγυήσει τελικά βγάζουμε εκτό παιδιά μια σειρά από παρόχου που δεν θα μπορούν να προσφέρουν τι επιλογέ αυτέ, γιατί είναι, θα είναι πολύ δύσκολο να το πράξουν. Και τρίτον, σε σχέση με τα τμήματα, με τα compartments είναι μήπως ε, γραφειοκρατική παραφροσύνη αυτή η πρόταση. Από τις παρατηρήσεις που έχω ακούσει από διάφορους ε, εκπροσώπους του κλάδου και ομιλητές σήμερα εδώ, παρανομιλητές τουλάχιστον, ε, μπορούμε να ζητήσουμε να θεσπιστεί αυτό ανατμήμα. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ερωτήσεις λοιπόν. Άρα από ένα λεπτό ο καθένας παρακαλώ για να απαντήσετε όλοι. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. για τα compartments, τα τμήματα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σίγουρα υπάρχουν περιφερειακές διαφοροποιήσεις. Το ΠΕΠ e δεν μπορεί να ε, προσφέρεται παντού στην Ευρώπη ε, χωρίς να υπάρχουν ε, θα υπάρχει περιφερειακή παροχή ασφάλισης αλλά όχι παντού. Πιστεύω ότι αν θέλουμε λύση για το ΠΕΠ, δεν πρέπει να συγχέουμε αυτό το θέμα με το IORP. Η ιδεώδης λύση είναι μία λύση όπου θα ε, δίνεται μια ε, επιδότηση. Το ΠΕΠ θα είναι συμπληρωματικό στη λύση του δεύτερου πυλώνα. Δεν θα αντικαταστήσει το δεύτερο πυλώνα. Ο, δεύτερο, ε, ο δεύτερος πυλώνας έχει κάποια όρια όμως. Γι' αυτό χρειάζεται να δούμε το ενδεχόμενο της συμπληρωματικότητας. Παρακαλώ. Ένα σχόλιο για τις εγγύησεις. Αν ρωτήσετε τους καταναλωτές και αυτοαπασχολούμενους, αρέσκονται στις εγγύησεις, αλλά εκεί δεν υπάρχει απόδοση. Υπάρχει γι' αυτό έλλειψη ασφάλειας. Ο συνδυασμός εγγυήσεων και κύκλου ζωής μπορεί να γίνει, αλλά οι εγγύησεις θα εισαχθούν αργότερα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο, γιατί υπάρχει διαφορά και στα βασικά εισοδήματα. Αν υπάρχει υψηλότερο βασικό εισόδημα, θα είναι λιγότερες οι εγγύησεις. Ε, ενώ ο κύκλος ζωής θα έπρεπε να έχει, έχει ε, ε, πιο μακρόχρονη βάση και έτσι εξασφαλίζεται απόδοση για την ερώτηση για το κύκλο ζωής και τις εγγύησεις. Ε, όπως είπαν από την Αμούντι, το 90% των προϊόντων κύκλου ζωής δίνουν καλό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, αν ε, κάνουμε μία ε, πρόβλεψη μπορούμε να πούμε ότι ε, απώλεια μπορεί να υπάρχει στον 1 στους 10 και μπορεί αυτή η απώλεια να πάει και μέχρι το 10 και το 20%. Στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ συνέβη αυτό στην οικονομική κρίση. Αν πούμε ότι κάθε ένα στους 10 μπορεί να είμαι εγώ και αν δέχομαι το 20% απώλειας του συνταξιοδοτικού μου εισοδήματος και απάντια είναι ναι, τότε η σωστή απάντηση είναι ο κύκλος ζωής. Συγκριτικά, η Solvency 2 ε, προβλέπει επίπεδο ασφάλειας ένα στα 200 χρόνια. Αν δηλαδή πάμε και ε, δούμε ποιος θα έχει απώλεια, μπορεί να είναι ένας στους 200 και αυτή θα είναι πολύ μικρότερη απώλεια από 10-20% δεν λέω ότι έχουμε τις δύο εναλλακτικέ, αλλά πρέπει να σκεφτούμε πολύ αν θα έχουμε ένα ΠΕΠ το οποίο θα έχει επίπεδο ασφάλειας και εγγύσεων και ποιότητας πανευρωπαϊκό και θα πρέπει να δούμε τι θα περιέχει αυτό. Μπορούμε να σκεφτούμε συνδυαστικά προϊόντα Μπορεί να υπάρχει δηλαδή ασφάλιση και διαχείριση ε, περιουσιακών στοιχείων. Να υπάρχει δηλαδή και το δεύτερο για να εξασφαλίζει μεγαλύτερη, υψηλότερη απόδοση. Η ΕΙΟΠΑ ε, λέει ναι στην πιστοποίηση, αλλά ε, επιμένει στην σωστή λύση στο θέμα των compartments, των τμήματων. Αντρέα Κοσολίνο, Σοσιαλιστές, Δημοκράτες. Ναι, αντικαταστώ τον κύριο Ατσόρου και θα σας διαβάσω το κείμενο που μου έστειλε και την ερώτησή του. Η πρόταση για την εισαγωγή ενός στεξωτικού πανευρωπαϊκού προϊόντος, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα από την εισηγήτρια στην εισαγωγική της παρέμβαση, είναι πολύ φιλόδοξη, ως προς την ουσία και ως προς το χρονοδιάγραμμα για να συμβάλλουμε στη λύση, στην αντιμετώπιση κάποιων από τις προκλήσεις που θα έχει τα επόμενα χρόνια η Ένωση να αντιμετωπίσει. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τον παραγόντα της δημογραφικής γύρανσης και μακροπρόθεσμα αυτό σημαίνει επιπλέον προκλήσεις και δυσκολίες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Επιπλέον ένα πανευρωπαϊκό συνταξιωτικό προϊόν μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην εξασφάλιση ε, αξιοπρεπούς επίπεδου σύνταξης για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, απέτηση μιας όλο και πιο κινητικής ε, εργατικής δύναμης. Θα πρέπει τα μέσα να είναι κατάλληλα για την εκμετώπιση των προκλήσεων και την πιο στενή ευρωπαϊκή ενοποίηση. Γνωρίζω ότι υπάρχουν στοιχεία στην πρόταση που χρειάζονται περαιτέρω διευκρίνηση, όπως άλλωστε προκύπτει και από τις συζητήσει, το φορολογικό, επί παραδείγματι, η φορολογική αντιμετώπιση αυτών των εξωτερικών προϊόντων, αλλά και η κατανομή σε διάφορα compartments και στις εξωτικές επενδύσεις. Και εν προκειμένου διατυπώνω την ερώτησή μου. Έγινε λόγος για την ε, default ε, εξορισμού δηλαδή επενδυτική σύνταξη τι θεωρούν οι προσκεκλημένοι μας απαραίτητο έτσι ώστε να υπάρξει επαρκής προστασία των καταναλωτών και πρόσβαση στην αγορά και για παρόχους που δεν θα είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή είναι η ερώτηση προς απευθύνει ο συνάδελφος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και ελπίζω η ανταλλαγή υπόψεων σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα να συνεχιστεί και να προσφέρει χρήσιμα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Μια συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν. Ποιος θέλει να αναλάβει την απάντηση. Παρακαλώ. για το πώς θα γίνει επιτυχές στο πρόγραμμα αυτό και για τους καταναλωτές. Το χαμηλό κόστος είναι σημαντικό. Αν είναι χαμηλό το κόστος τότε έχουν περισσότερα κέρδη στο χαρτοφυλάκιό τους οι ίδιοι οι επενδυτές. Τώρα για την πρόσβαση των μικρών παρόχων έτσι ώστε να υπάρχει ισότητα στην αντιμετώπιση μικρών και μεγάλων. Το θέμα είναι ακριβώς ποια είναι τα φορολογικά καθεστώτα στα διάφορα κράτη-μέλη και εδώ η ΑΙΟΠΑ θα μπορούσε να βοηθήσει και τους μικρούς παρόχους να λειτουργήσουν σε πολλές χώρες. Θέλετε κι εσείς να απαντήσετε, η κυρία Φίλη. Το θέμα του κόστους είναι κάτι το οποίο είπε ο συνάδελφος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσύ, εμείς είμαστε υπέρ του μεγάλου αριθμού των παρόχων και επίσης είμαστε υπέρ των συμβολέων τα οποία μπορούν να γίνουν ε, διαδικτυακά εδώ θα μπορούσαμε ε, να ενημερώνουμε κάπως καλύτερα τους καταναλωτές στην επιλογή τους. Δεν μπορώ να κάνω βέβαια εδώ συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ε, δυνατότητες. Ε, η στρατηγική του κύκλου ζωής όταν εφαρμόζεται σωστά είναι κάτι το οποίο μπορεί να ληφθεί πραγματικά υπόψη. Λοιπόν, από τους συντηρητικούς δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή εδώ. Οπότε θα περάσω στον εκπρόσωπο της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες προοπτικές για το ΠΕΠ που αρουσίασαν. Το θετικό είναι ότι φαίνονται τα διαφορετικά συμφέροντα ε, στον κλάδο. Η ομάδα μου δεν θα σας εκπλήσει ότι έχει μια σοβαρή επιφύλαξη απέναντι σε τέτοια ιδιωτικά προϊόντα. Θα έπρεπε να υπήρχε αξιοπρεπής ε, συνταξιοδότηση η πρόσφατη πολιτική εμπειρία της χρηματοπιστωτικής κρίσης και στις Ηνωμένε Πολιτείες αρχικά ε, είδαμε ότι ε, είχε καταστροφικά αποτελέσματα, άνθρωποι έμειναν χωρίς σύνταξη, αλλά και στη γερμανική αγορά όπου εισαγάγαμε τη λεγόμενη σύνταξη Ρίστερ, ένα προϊόν το οποίο δεν ε, εξελίχθηκε καλά, ίσως ε, θα υπάρξουν και αντιρρήσεις εδώ, αλλά νομίζω ότι και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση επέκρινε το πρόγραμμα Ρίστερ για τις συντάξεις. Ε, είχε συμβάλει τότε το προϊόν αυτό στη μείωση των συντάξεων και στην ανάγκη συμπληρωματικών ε, συντάξεων. Υπάρχει κάποια μελέτη που δείχνει ότι με το ΠΕΠ ε, ε, περίπου 700 δις θα περάσουν σε αυτή την αγορά. Από πού θα προέλθουν τα χρήματα αυτά. Είναι ιδιωτικές αποταμιεύσεις. Και μία δεύτερη ερώτηση στην κυρία Φιλή. Τι ωφέλη βλέπετε ε, για την προστασία των ε, καταναλωτών. Πόσο θα προστατεύσει το προϊόν αυτό σε σύγκριση με άλλα ε, συνταξιοδοτικά προγράμματα αναδιανεμητικά. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις έγιναν. Η πρώτη νομίζω για τον Τομπία Σεμπίχλερ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Δεν ξέρω από πού προέρχονται τα 700 δις στη μελέτη. Εγώ προσωπικά πιστεύω όταν μιλάμε για πολιετή ορίζοντα, αναπόφευκτα θα αρχίσουμε με πολύ χαμηλότερα ποσά. Δεν γνωρίζω ακριβώς πού βρήκατε τον αριθμό στον οποίο αναφερθήκατε. 700 δις καταθέσεων. Να πούμε ότι τέτοιου είδους συνταξιοδοτικές λύσεις δεν ε, θα χρησιμοποιούν χρήματα μόνο από αυτού του είδους την αποταμίευση. Ε, θα χρηματοδοτούνται από την αγορά, θα προσπαθήσουν να γίνουν κατανοητά στην αγορά ως εκ τούτου ελκυστικά και νομίζουμε ότι μέσω πρόθεσμα τουλάχιστον θα υπάρξει δυνατότητα παροχής μιας σωστής λύσης, συμπληρωματικής λύσης εμείς δεν θέλουμε να αποσυρθούν οι αποταμιεύσεις από τα υπάρχοντα συνταξιοδοτικά συστήματα. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Και δεν θα πρέπει να είμαστε σε ανταγωνισμό με τα εθνικά συνταξιοδοτικά προγράμματα τα οποία είναι, προτείνονται στις αγορές. Και μία ερώτηση για την κυρία Φίλη. Δεν ξέρω, υπάρχουν εκπρόσωποι και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θέλουν να μιλήσουν για τα 700 δις και τα λοιπά. Όπως είπα στην παρουσίασή μου, το ΠΕΠ δεν είναι το μαγικό όπλο για να λυθούν τα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε σε συνταξιοδοτικό επίπεδο. Τα βασικά καλά χαρακτηριστικά των ΠΕΠΣ είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στον τομέα των συντάξεων και να υπάρξει δυνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα στους πολίτες, αλλά σίγουρα δεν είναι μία μαγική λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τώρα για το θέμα των 700 δις Επιτροπή για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που θέσατε την ερώτηση αυτή. Οι αριθμοί α, τους οποίους αναφέρατε προέρχονται από την εκτίμηση επιπτώσεων η οποία συνοδεύει την πρότασή μας. Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, ε, το προϊόν αυτό θα συνεισφέρει στο να αντιμετωπιστεί το κενό που υπάρχει ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα συντάξεων. Θα βοηθήσει όμως. Είναι σαφές ότι πολλοί καταναλωτές ε, έχουν προβλήματα λόγω της έλλειψης προσφορών. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε μία δημόσια διαβούλευση και ακριβώς ε, είχαμε 500 απαντήσεις που ανταποκρίθηκαν στα ερωτήματά μας ε, σε προσωπικό επίπεδο για τα σχόλιά τους ε, σε σχέση με το επίπεδο της, των μέσων και των επιλογών τα οποία είχαν στη διάθεσή τους, ε, το σύνδρομο αποκλεισμού, ε, ο ανεπαρκής αριθμός προσφοράς και η έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με τον καθορισμό των ασφαλίστρων. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε εμείς κάνοντας μία πρόταση για ένα συμπληρωματικό μέσο εθελοντικού χαρακτήρα που θα επιτρέψει σε ορισμένους που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους προσωπικές συντάξεις ή επαγγελματικές συντάξεις να το κάνουν. Αυτό απασχολούμενοι σαν παράδειγμα που δεν μπορούν να συνεισφέρουν σε ένα IORP σύμφωνα, σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα. Θα μπορούν να το κάνουν με τα PEP e Επίσης και για θέματα όπως ε, ε, το, τα προβλήματα ανάμεσα στα φύλλα, οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα. Μία μητέρα η οποία για λόγους πρακτικούς δεν μπόρεσε να συνεισφέρει σε επαγγελματικά προγράμματα για διάφορα χρόνια και θα μπορεί να συνεισφέρει συμπληρωματικά σήμερα σε ένα ΠΕΠ. Πήραμε στοιχεία από την αγορά και πήραμε και γνωμοδοτήσεις από πλευράς της ΕΙΟΠΑ. Και η πρόβλεψη λέγει ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο προσωπικών συντάξεων που να φτάνει πράγματι σε 2.100 δις με κίνητρα φορολογικά από διαφορετικές πηγές. θα υπάρξει καταρχάς μια πραγματική και γνήσια ενιαία αγορά. Η αγορά σήμερα για προσωπικές συντάξεις είναι πολύ διασπασμένη. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ανοιχτή αγορά. Θέλουμε να ανοίξουμε περισσότερο τον αριθμό των παρόχων που θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τέτοια προγράμματα. Θα υπάρχουν λοιπόν περισσότερα προγράμματα και ελπίζω και καλύτερα προγράμματα γιατί θα υπάρξει αυξημένος ανταγωνισμός αυτοί που δεν έχουν αρκετή παροχή ε, προϊόντων θα είναι σε θέση μέσω των ΠΕΠ να συνεισφέρουν. Και νομίζω ότι θα αυξήσουμε τις εμπορικές ε, πρόσφορες που θα επιτρέψουν ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι έχουν χαμηλά έσοδα να συνεισφέρουν με χαμηλά ε, επίπεδα συμμετοχής. Τώρα για τα φορολογικά κίνητρα και αυτό είναι ένα σημαντικό ε, θέμα. Η αύξηση σαν παράδειγμα του επίπεδου των εθνικών συντάξεων είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει στο ποσό αυτό στο οποίο εμείς αναφέρουμε τα 2.100 δις. Λοιπόν, περνάμε στον επόμενο σκιώδη, Άνεμανς, ENF. Πρόεδρε, έχω μια πολύ στενή ερώτηση να διατυπώσω στον καθηγητή Βαν Μέρτεν για τον τρίτο πυλώνα που προτείνεται. Γιατί στο Βέλιο, παραδείγματι, θα ήταν ανταγωνιστικό για τα συνταξιωτικά ταμεία που ε, χαίρουν ενός ευνοϊκού φορολογικού συστήματος. Θα εσύ αυτό και για το ΠΕΠ αντίστοιχα. Έτσι θα είναι, θα είναι συμπληρωματικό. Αλλά τότε δεν υπάρχει ο κίνδυνος ε, να αποχωρήσουν από τα εθνικά συστήματα σταξιδότησης ε, οι συντάξεις και βέβαια και τα σχετικά κονδύλια. Απάντηση. Πριν απαντήσω στην ερώτηση αυτή, κύριε Χέις, δεν σκόπευα να επικρίνω τα θετικά της οδηγίας ΣΥΟΡ 2 που υπάρχουν. Απλώς σημειώνω ως ειδικό και σε σχέση με την ΕΡΟΠ, ενώ ότι πρέπει να εξυπηρετηθεί ο στόχος της καλύτερης διακίνησης. Ιδιαίτερα στα, όντιση, στα σαφώς προσδιορισμένα συστήματα εισφορών. Το πλεονέκτημα από την ΕΟΡΠ δεν το βλέπω. Αυτό είχα να πω. Τώρα η άλλη ερώτηση ήταν εάν ένα ΠΕΠ θα μπορούσε να επηρεάσει το φορολογικό σύστημα του δεύτερου πυλώνα. Σας κατάλαβα καλά. Όχι, τα χρήματα που θα αποχωρήσουν ε, από τα εξωτικά ταμεία. Πάντα λέω και ναι και ου. Ναι, διότι βεβαίως για τις κατοχώρες όταν ε, η εξαίρεση του τρίτου πυλώνα εξαρτάται από τις επιλογές για τον πρώτο και δεύτερο, ότι η απάντηση μπορεί να είναι καταφατική. Αλλά το ίδιο σύστημα δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες και άρα δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει στο Βέλγιο. Και προσπαθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εγκαθιδρύσουμε αυτό το σύστημα των αντισταθμίσεων, σταδιακών αντισταθμίσεων. Αλλά υπάρχουν και κράτη-μέλη στα οποία δεν ισχύει το σύστημα αυτό και άρα εκεί δεν θα υπάρχει τέτοιο, τέτοια συνέπεια για τα εθνικά συνταξιδοτικά συστήματα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε και το γύρο των σκιωδών. Έχουμε όμω και δύο ε, επιτροπές με γνωμοδότηση. Από την Επιτροπή της Απασχόλησης, κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ καταρχάς που μας έδωσε την ευκαιρία για αυτή την ακρόαση. Έρχομαι εδώ για να μάθω, έτσι πιστεύω, γιατί εγώ την έκθεση την ε, εξετάζω από μια άλλη σκοπιά, πολιτική σκοπιά, με καθήκον πάνω απ' όλα προσέγγιση την απασχόληση εκ μέρους Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι σαφή η εντολή μου και νομίζω ότι το ΠΕΠ θα πρέπει απολύτω ξεκάθαρα να είναι συμπληρωματικό και να μην αναμεικνύεται με το δεύτερο πυλώνα πρώτα απ' όλα, αλλά ούτε και με τον πρώτο, με το συμπάθειο. Και έτσι θέλω σαφή τοποθέτηση σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Τη βλέπω θετικά, ελπίζω και ο κλάδος με τους ε, επιφανείς εκπροσώπους του που έχουμε εδώ να δει όχι τα προβλήματα αλλά τις λύσεις αυτών περισσότερο γιατί ένα τέτοιο προϊόν θα μπορούσε να καταστεί ιδιαίτερα ελκυστικό ευρωπαϊκό προϊόν και ξέρετε σε ε, πόση ανάγκη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, τονώσει το κύρος της και την εικόνα της σε σχέση με τα προϊόντα που προσφέρει στον πολίτη. Γι' αυτό και πιεζόμαστε και χρονικά σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Αυτό που θα ονόμαζα πολιτικό μάρκετινγκ το προφανές λέω, αλλά ας είμαστε και προσεκτικοί, διότι απευθυνόμαστε εδώ σε ομάδες στόχους, το είπε ευτυχώ και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ίδια. Και βλέπω ότι έχω πολλά ακόμα να μάθω, επί παραδείγματι. Υπάρχουν γονείς που θέλουν να κάνουν ένα τέτοιο δώρο στα παιδιά τους. Ε, αν η επένδυση είναι ε, τον 50 ευρώ μέσα σε κάποιες δεκαετίες προσφέρει ένα εξαιρετικό προϊόν και όταν έρθει η ώρα ο νέος αναλαμβάνοντας και μια θέση εργασίας να αναλάβει και τη σχετική καταβολή των εισφορών τότε έχουμε ένα τεράστιο έργο για την Ευρώπη, για την Ενωμένη Ευρώπη και πρέπει να το υποστηρίξουμε με θετικό τρόπο. Και γι' αυτό ιδιαίτερα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ θέλω να πω ότι έχει τις αρμοδιότητες, είναι οι προσπάθειες θετικές, είναι ιδιαίτερος ικανή η συγγητριά μας και εγώ εκ μέρους της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων θα προσπαθήσω να συμβάλλω με κάποιες διαφορετικές ιδέες ή μια διαφορετική θεώρηση, αλλά πάντως όχι με αντίδραση, με αντίθετες θέσεις. Ευχαριστώ πολύ και κυρία από την ΕΜΚΟ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή για την ακρόαση που ήταν ενδιαφέρουσα. Αν και τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν και άλλες ερωτήσεις. Εγώ επικεντρώνομαι στην προστασία των καταναλωτών και το ΠΕΠ θα είναι πιο επιτυχημένο από άλλα προϊόντα θα πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής από πριν τι θα κερδίσει για να μπορεί να συγκρίνει με άλλα εθνικά προϊόντα που ίσως είναι περισσότερο ή λιγότερο καλά. Υπάρχει και το ευρωπαϊκό επίπεδο που περιπλέκει τα πράγματα. Ας πούμε το παράδειγμα των compartments. Παράδειγμα, είτε στη Γερμανία είτε στη Γαλλία, δεν έχει σημασία, ε, ε, δίνετε στις εισφορές σας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν αλλάξετε υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ε, αν ε, το βλέπω σωστά, στη Γερμανία το όριο ηλικίας είναι 67, σε άλλες χώρες είναι 65 κλπ. Τι ισχύει. Δεν έχουμε εναρμονισμένα φορολογικά συστήματα. Ε, πώς φορολογούνται οι συντάξεις με διαφορετικό τρόπο. Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν το σύστημα αν κάποια στιγμή θέλει κανείς να συγχωνεύσει το μίση ή ε, σε κάποιο χώρα μπορεί να ε, ισχύει ηλικία συνταξιοδότηση 62, άλλους 67. Πώς θα γίνουν οι υπολογισμοί. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες της Κομισιόν Εμάς μας ενδιαφέρει ένα καλό, διαφανές προϊόν για τον καταναλωτή. Ε, θα πρέπει να είναι ενημερωμένος ο καταναλωτής. Θα πρέπει να μην είναι πολύ δαπανηρό και να εξαφανίζονται ε, οι αποταμιεύσεις τους σε επιβαρύνσεις. Να είναι ένα καλό προϊόν. Αυτό θέλουμε. Ε, η ιδέα του ΠΕΠ είναι καλή, αλλά πρέπει να υπάρξουν κάποιες διευκρινήσεις γιατί πολλά ζητήματα είναι ακόμα ανοιχτά. Ευχαριστώ πολύ για τη δήλωση. Δεν βλέπω κανέναν στη διαδικασία του Catch the Eye. Α, υπάρχει. Η κυρία Περές. Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων Το χρονοδιάγραμμα είναι φιλόδοξο, αλλά θα το συζητάμε το θέμα αυτό για πολύ καιρό. Ζητώ συγγνώμη από τους δύο ομιλητές που δεν άκουσα, αλλά σχετικά με τη φορολογία, από αυτά τα οποία άκουσα, είναι προφανώς ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε κάθε φορά όταν έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίε των χρηματαγορών ε, θέλουν τη δημιουργία ενός διασύνοριακού προϊόντος στο οποίο να συμμετέχουν ε, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και πολίτες ε, χωρίς καμία δυσκολία και τίθεται το θέμα ενός φορολογικού καθεστώτος το οποίο να καλύπτει αυτές τις δυνατότητες σχετικά με την, δυνατότητα μεταφοράς. Δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι ε, το προϊόν αυτό δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς όνει και καλά. Δεν λύνει ε, θα έλεγα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα στους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, ανοίγει μια πόρτα αλλά θα πρέπει τα υπάρχοντα καθεστώτα να γίνουν πιο μεταφέρσιμα σε εισαγωγικά. Τώρα για την fallback option έχω την αίσθηση ότι επί της αρχής ε, συμφωνούμε. Θα πρέπει όμως να υπαλληθεύσουμε με τους προσκεκλημένους και θα θέσω το θέμα σε όλους τους εμπειρογνώμονες να αναγνωρίσουν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικό συνταξιοδοτικό προϊόν. Οπότε η default option θα πρέπει να είναι πάντα συνταξιοδοτική λύση και προϊόν και όχι επενδυτικό γενικότερα. Και θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις πέραν της ονομαστικής απόδοσης αν θέλουμε το προϊόν αυτό να είναι πράγματι ελκυστικό. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά αυτά ήταν τα θέματα πάνω στα οποία ήθελα να σταθώ. Μια τελευταία παρατήρηση για την ΑΙΟΠΑ. Για την ΑΙΟΠΑ τέθηκε το θέμα από πολλούς ομιλητές. Η μεταρρύθμιση η οποία προτείνεται στην παρούσα φάση καλύπτει υποτίθεται τις ανησυχίες σας ή μήπως πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Έχουμε 10 λεπτά τώρα για να κλείσουμε τη συζήτηση. Να ζητήσω λοιπόν από τους ομιλητές μας να μας πούν τρεις-τέσσερις τελευταίες φράσεις απαντώντας και στις ε, ερωτήσεις της κυρίας Μπερές και των προηγούμενων ομιλητών. Και μετά να δώσουμε το λόγο στην Σοφή για να κλείσει. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την ανάποδη σειρά. Θα συμφωνήσω μαζί σας, λέει ο κύριο Έρλεμενς, ότι το προϊόν αυτό θα πρέπει να είναι ένα συνταξιοδοτικό προϊόν, όχι ένα προϊόν κεφαλαίου αποκλειστικά. Και αυτό θα εξαρτηθεί από τα καθεστώτα τα διάφορα που ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και ακριβώς οι πληροφορίες οι οποίες θα μπορεί να δοθούν θα κρίνουν την επιλογή αυτού του προϊόντος από άλλα προϊόντα που ε, στοχεύουν ε, στην αύξηση των κερδών μέσω αύξηση κεφαλαίων. Έχουμε ένα πρόβλημα χρόνου. Μια στιγμή, παρακαλώ να τους δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να απαντήσουν και αμέσως μετά θα σας δώσω το λόγο. Η κυρία Φίλη. Για να απαντήσω στην κυρία Μπερές. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχει την ε, επιλογή ο καταναλωτής. Έχει διαφορά βέβαια η καθεθνική νομοθεσία. Μερικές φορές προτιμάται ε, η σύνταξη, άλλες φορές ε, κατά κεφάλαιο ή ο συνδυασμός αυτών. Πάντως πρέπει να μείνει στον καταναλωτή η επιλογή. Για τη μεταρρύθμιση των εποπτικών αρχών δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι, διότι η προστασία των καταναλωτών δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ως πτυχή στη μεταρρύθμιση αυτή. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θεωρούμε ότι είναι καλό το σύστημα πιστοποίησης των ΠΕΠ της ΑΙΟΠΑ. Φαρμίρε, Φανμέρτεν. Λίγες ε, παρατηρήσεις ε, για τα compartments και τη μεταφορικότητα. Δεν λέω ότι λύνει όλα τα προβλήματα. Αλλά η προσέγγιση κατά τμήματα είναι πολύ πρωτότυπη. Ενισχύει τη δυνατότητα μεταφοράς, περαιτέρω, χωρίς να είναι τέλεια. Δεν θέλω να επενεχθώ κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ένα ή θα ήταν ακόμη καλύτερο. Και σταματώ εδώ. Ο επόμενος ομιλητής παρακαλώ, ο κύριος Δεν ε, θα συνεχίσω στο επιχείρημα αυτό, διότι εκπροσωπώ τους καταναλωτές και έχω τελείως διαφορετική άποψη αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή για να μιλήσουμε για το θέμα. Είχα την ελπίδα πως θα μπορούσαμε να βρούμε μια καλή λύση που δεν θα επιβληθεί όμως τα κρατη αλλά που θα ήταν προτιμότερη για να διευκολύνεται η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων που είναι και το κλειδί όλης αυτής της ε, επιχείρησης. Ευχαριστώ κύριο Σμπίρχιλερ. Ναι, όντω για μα είναι η φορολογία το κλειδί. Καλή λύση δεν έχουμε. Είμαστε τεθειμένοι σε καλή συνεργασία, σε υποδομητική συνεργασία με του πάντες για να βρούμε μια καλή λύση. Ε, πάλι ερχόμαστε στο θέμα των τμήματων, των compartments. Εάν υπάρχουν ε, τα compartments, αν διατηρηθούν δηλαδή, μιλούμε για εθνικέ λύσει, αν μιλούμε για ε, πανευρωπαϊκό προϊόν υπό το καθεστώ τη δεύτερη ΙΟΡΠ, τότε η ΟΠΑ μπορεί να δραματίσει το ρόλο τη. Ευχαριστώ πολύ. Σοφίνη Φέλτ, συγκεκριμένη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ομιλητές και τους συναδέλφους για την συνεισφορά τους. Δεν θα κάνω καθόλου δηλώσεις για να μην ενοχλήσω ή φοβήσω κανέναν. Θα προχωρήσω με σταδιακά, θα γίνουν περισσότερες διαβουλεύσεις που θα ενταχθούν στα έγγραφα εργασίας μας. Ε, θα παρουσιάσω τον Ιανουάριο. Μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Προς τον συνάδελφο από την ΚΟΕ. Καταλαβαίνω αυτό που είπατε, αλλά εδώ μιλάμε για πρόσθετο συμπληρωματικό σύστημα. Κι αν στα κράτη-μέλη το κράτος δεν επαρκεί, αυτό δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη, έχει να κάνει με τις εθνικές αρχές που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Αν θα είναι το ΠΕΠ συμπληρωματικό, θα είναι συμπληρωματικό προς κάτι. Και αυτό είναι το καθήκον των εθνικών αρχών, όπως προβλέπουν οι συνθήκες. Δεν είναι μόνο αρμοδιότητα, είναι και καθήκον τους. Δεύτερον, και αυτό συνδέεται με τις ε, παρατηρήσεις ε, του κ. Άλμανς και άλλων. Υπάρχουν ανησυχίες στα κράτη-μέλη. Βεβαίως θα ήταν πολύ αστείο να έχουμε ένα σύστημα που θα επηρέαζε αρνητικά ή θα υπονόμευε τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα, κυρίως εκείνα που είναι καταξιωμένα και στιβαρά. Δεν θα το κάναμε αυτό ποτέ. Υπάρχουν πολλοί που εξετάζουν το φάκελο και κάποιος θα, ε, είναι βέβαιο ότι θα εντοπιστούν ε, τέτοιου είδους προβλήματα. Ε, πρέπει λοιπόν να είναι συμπληρωματικό. Όμως υπάρχει ένα κενό συνταξιοδοτικό. Σε κάποια κράτη οι συντάξει είναι πολύ καλές, όχι τέλειες, ακόμα και στη δική μου τη χώρα, την Ολλανδία, όπου έχουμε ένα πολύ στέρεο σύστημα και αυτό όμως πρέπει να προσαρμόζεται στις αλλαγές στην κοινωνία, την αγορά εργασίας, στις δημογραφικές αλλαγές, χρηματοοικονομικές αγορές κλπ. Το σύστημα θα μεταρρυθμιστεί και εκείνο. Ε, ε επίσης ε, μιλήσατε και για την ε, διαφορά στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών χαμηλότερες για τις γυναίκες που πρέπει να αποταμιεύουν περισσότερο για να φροντίζουν το συνταξιοδοτικό τους. Τώρα, η φορολογική αντιμετώπιση. Αυτό είναι πολύ λεπτό αλλά και σύνθετο ζήτημα. Νομίζω ήταν σωστό από πλευράς Κομισιόν να μην ενταχθεί στον κανονισμό αλλά να γίνει χωριστή σύσταση γιατί θα ήταν αυταπάτη να πιστέψουμε ότι θα υπήρχε κάποια ομοφωνία σε αυτό το θέμα για να μην μιλήσω για συνένεση. Όμως θεωρώ ότι μπορούμε να συζητήσουμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και να βρούμε τρόπους για να επεξεργαστούμε την σύσταση της Κομισιόν και να δούμε μήπως μπορούμε να βρούμε μια σύσταση που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη σε βάση προαιρετική να προχωρήσουν σε κάποια εναρμόνιση. Ίσως αυτός θα ήταν ένας τρόπος για να προχωρήσουμε εδώ. Και βέβαια σε τελευταία ανάλυση, όπως και αν είναι το ΠΕΠ, πρέπει να τύχει της εμπιστοσύνης των ε, πολιτών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι κάτι καινούριο, δεν είναι γνωστό δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό, οπότε θα το δούνε με κάποια δυσπιστία και αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε, να είναι και ελκυστικό και για τους παρόχους, γιατί αν δεν είναι ελκυστικό δεν είναι επιχειρηματικό προϊόν και δεν έχει νόημα να το συνεχίζουμε. Τώρα για τα compartments, για αυτά τα τμήματα, τα επιμέρους ή τους τομείς πρέπει να βρεθεί λύση. Νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν ότι ο πάροχος θα πρέπει να έχει τμήματα μέσα σε πέντε χρόνια σε κάθε κράτος μέλος δεν είναι εφικτό. Πρέπει να βρεθεί άλλη λύση. Ίσως γιατί οι μικροί πάροχοι, οι περιφερειακοί θα υποστούν διακρίσεις αρνητικές ή μπορεί να υπάρξουν και κάποιες ρυθμίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Η ΕΙΟΠΑ εδώ μπορεί να τα διευκολύνει αυτά. Και τέλος, για το IORP. Στη χώρα μου υπάρχει μεγάλη ευαισθησία και ο κύριος Χάνεμαν το είπε. Βέβαια, αν έχουμε ένα σύστημα με το IORP που λειτουργεί καλά, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην το υποσκάψουμε. Να πούμε, τα IORP εξαιρούνται. Δεν ξέρω αν αυτή η ριζική λύση είναι η καλύτερη. Υπάρχουν και ενδιάμεσες λύσεις που δεν θα επηρεάσουν αντικά τα υφιστάμενα συστήματα, τα εθνικά, και, και κάποιες άιορψε, ε, κάποιες κατηγορίες άιορψε, δηλαδή ε, στα εξαιρετικά σχέδια. Ο κύριος Άρλιμανς νομίζω το είπε αυτό. Ε, μίλησε για κατανομή μέσω άλλων νομίμων μέσων. Εγώ είμαι πολύ ανοιχτή σε αυτό. και θα κάνω διαβουλεύσεις και με πολλούς ανθρώπους τις επόμενες εβδομάδες και θα σας υποβάλω τον Ιανουάριο το έγγραφο εργασίας μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σε καλά χέρια λοιπόν η έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν και τους σκιώδεις εισηγητές και φυσικά τους προσκεκλημένους μας. Η επόμενη ανταλλαγή απόψεων θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 25 Μαρτίου, εξέταση τροπολογιών 23-24 Απριλίου και 4 Ιουνίου θα ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την εκκίνηση της διαδικασίας, σας ευχαριστώ όλους και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως.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 Παρακαλώ. Περάστε στις θέσεις σας για να ξεκινήσουμε το δεύτερο θέμα της απόψινής συνεδρίασης. Και όσοι θέλετε θεμερίες επαφές ακόμη, παρακαλώ, εκτός αιθούσης για να συνεχίσουμε. Uh, Οδηγία για την ε, παροχή αρμοδιοτήτων στι αρχέ ανταγωνισμού των κρατών μερών ώστε να του κανόνε για τη διασφάλιση εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Και παρακαλώ όποιος δεν θέλει να λάβει μέρος στη συζήτηση αυτού του τμήματος, του θέματος, να αποχωρήσει από την αίθουσα. Πάνω από 250 τροπολογίες για την πρόταση αυτή με τις ελάχιστες ε, προδιαγραφές και εγγύησεις. που επιτρέπει στις εθνικές αρχές να αναπτύξουν το δυναμικό τους, ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση της ε, κατάχρησης της πόσουσας θέσης θα πρέπει τα κρατη να εφαρμόζουν τις ίδιους κανόνες. Και το Συμβούλιο επεξεργάζεται τη νομοθετική πρόταση. Η Εστονική Προεδρία έχει ξεκινήσει τη δουλειά που θα συνεχίσει η Βουλγαρική κατά πάσα πιθανότητα για το δεύτερο τριμηνό του 18 και ο εισηγητής για το λόγο αυτό προτείνει να αναβάλουμε έως τα τέλη Φεβρουαρίου την ψηφοφορία του σχεδίου στην ΕΚΟΝ για να έχουμε περισσότερο περιθώριο για συμβαστικές τροπολογίες τον εισηγητή Σήμερα καθιστά ο κύριος, η κυρία Σάντερ. Εισηγητής Σκιώδης έκαστος από πέντε λεπτά και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού άλλα πέντε. Πρόεδρε, κυρία Σάντερ, αγαπητοί συνάδελφοι, στα αγγλικά. Θα ήθελα να στείλω συγγνώμη εκ μέρους του του κυρίου Σβάμπο, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα και με παρακάλεσε να σας προσώσω τα εξή σχόλια. Ο εισηγητής θέλει να ευχαριστήσει τους και όδης εισηγητές και όλους τους άλλους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες και ως εκ τούτου προσέφεραν τα μάλα για τις διαπραγματεύσεις στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Σφάμπ πιστεύει ότι οι τροπολογίες αυτές αποτελούν καλή βάση για επικοδομητική συνεργασία και συμβασμούς. Αρκετές τροπολογίες ακολουθούν ε, τους ίδιους στόχους και ως εκ τούτου θεωρεί ότι μπορεί τουλάχιστον για ορισμένα άρθρα να βρεθεί εύκολα συμφωνία. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει προσαρμογή και να αποσταλεί το ταχύτερο ε, το κείμενο για να μην επισέλθουμε σε υπερβολικά και πολλές λεπτομέρειες. Σήμερα ο εισηγητής θέλει να επισημάνει μόνο λίγα σημεία. Πρώτον, χέρι ο εισηγητής που όλες οι ομάδες συμφωνούν πως χρειάζονται ελάχιστες προδιαγραφές και εγγύησεις προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική επιβολή των κανόνων για τον ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ως εκ τούτου είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία στη διάθεσή τους για την επιβολή των κανόνων για, την, για τον ανταγωνισμό. Ε, διασφαλιστική δικλίδα άρθρου 3, όπως αναφέρθηκε και, στο σχέδιο, ε, είναι καλή ιδέα, ωστόσο πιστεύει ο εισηγητής ότι η ενίσχυση των ε, αρμοδιοτήτων επιβολής πρέπει να ισοσταθμίζεται από διαδικαστικές εγγυήσεις, δικονομικές εγγυήσεις και, ε, και παραπέμπει στον θεμελιώδη χάρτη αλλά και τη γενική και λέει ότι ο θεμελιώδης χάρτης και η παραπομπή στις γενικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αρκούν και άρα θα πρέπει να υπάρχουν οι διασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου να ε, καλυφθούν οι διαδικασίες των άρθρων 101 και 102 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητής χαίρεται που συμφωνούν και οι άλλοι και οι σκιώδες δηλαδή και έχουν υποβάλει αντίστοιχε τροπολογίες. Άρθρο 11 και υποχρεώσεις. Χαίρεται ο εισηγητής επίσης γιατί βλέπει ότι υπάρχει συμφωνία ως προς την ε, χρήση των αποφάσεων για τις υποχρεώσεις που επανακινούν τις διαδικασίες κυρίως σε περιπτώσεις όπου παραδείγματι μπορεί να έχει ε, υπησέλθει ουσιαστική αλλαγή ή σε περιπτώσεις όπου μια απόφαση έχει ληφθεί μένα αλλά οι επιχειρήσεις ε, αναλαμβάνουν δράση αντιθέτη με τις δεσμεύσεις της υποχρεώσεις τους. Άρθρο 14. Και πρόστιμο. Υπάρχει ένα ανατατόριο. Ωστόσο, φαίνεται εδώ να εκφράζονται αποκλίνουσες απόψεις για το πώς αυτό μπορεί να επιβάλλεται. Και ο εισηγητής θεωρεί ότι αφού πρώτα σε πρακτικούς όρους τα κράτη-μέλη έχουν στο σύνολό τους ήδη προβλέψει το 10% του κύκλου εργασιών ως μέγιστο πρόστιμο και δεύτερον οι αρχές εφαρμόζουν τα άρθρα 101 και 102 όπως άλλωστε και η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσετε το ίδιο το πρόστιμο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προς το στόχο και μιας πιο ομοιόμορφης προσέγγισης αλλά και ενός πιο προβλέψιμου συστήματος. Εάν ξεπερνάει το 10% ένα μέγιστο πρόστιμο θα είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα συνήθη παράνομα κέρδη ε, που προκύπτουν από την παραβίαση των κανόνων για τον ανταγωνισμό. Επίοικια. Ο εισηγητής με ικανοποίηση σημειώνει ότι κάποιες τροπολογίες που προτάθηκαν ζητούν πιο αποτελεσματικά προγράμματα επίοικιας ε, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την ασφαλεία δικαίου, για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να οθούνται και αυτές να συνεργάζονται με τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές και επίσης πρέπει οι αποκλήσεις μεταξύ εθνικών συστημάτων επί, επίοικιας να μειωθούν Θα πρέπει δηλαδή να είναι οι ίδιοι όροι από του οποίου θα δίνεται είτε απαλλαγή είτε μείωση προστήμου από τις εθνικές αρχές. Ο εισηγητή προσβλέπει σε μια επικοδομητική συνεργασία με τους Κιώδης τις επόμενες εβδομάδες. Και... Ενημερώνει, όπως είπατε άλλωστε και εσείς, ότι τα προβλήματα στην πληροφορική που αντιμετωπίσαμε οδήγησαν σε αναβολή της προθεσμίας, σε παράταση προθεσίας για, τις προθεσμίες για την κάθε τροπολογιών έως 27 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την αντικατάσταση ε, του εισηγητή. Τι Μπορτσάνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. λόγω των προβλημάτων ε, σε επίπεδο πληροφορικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έπρεπε να αναθεωρήσουμε όλες τις συναντήσεις μας στο χρονοδιάγραμμα. Πάντως ο εισηγητής λειτουργεί επικοδομητικά και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας μαζί του και στο μέλλον. Να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θα θέλαμε να έχει η παρούσα πρόταση. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι η ανεξαρτησία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού πρέπει να είναι δεδομένη. Όχι μόνο μέσω των κανόνων και να μην επιτρέπεται η αντικατάσταση των ηγετικών ομάδων των υπηρεσιών, αλλά και η δυνατότητα να λειτουργήσουν με λειτουργικό τρόπο. Δεύτερον, η όθηση που θα δώσουν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού πρέπει να συνοδεύονται από την κατάλληλη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να υπάρξει προσοχή στο πώς χρησιμοποιείται ε, η πίστοση την οποία έχουν στην διάθεσή τους οι υπηρεσίες αυτές. Τρίτον, να υπογραμμίσω ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια. Οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες έχουν ανάγκη από σωστή ενημέρωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να είναι σε θέση να αναγυγνώσκει τις ετήσιες εκθέσεις όλων των αρχών επί του ανταγωνισμού. και θα πρέπει να έχουμε στην διάθεσή μας και τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες αυτές μέσω iCloud και τα λοιπά. Να επαναλάβω για μια ακόμη φορά τη διαφορά ανάμεσα στα προσβάσιμα θεωρητικά στοιχεία και στα στοιχεία τα οποία έχει κανείς στη διάθεσή του όπως επίσης και την διαφορά ανάμεσα στις έννοιες του σχετικού και του μη σχετικού γύρω από τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες αυτές. Σας ευχαριστώ για την ομάδα των συντηρητικών ο κύριος Ταρμπάτη. Ε, εμείς συμφωνούμε με την έκθεση ΣΟΑΜ. είναι πολύ σημαντική έκθεση. Οι δυνατότητες ε, ελέγχου νομίζω κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Στη τελευταία ακρόαση με τις αρχές ε, για τα καρτέλ ε, έδωσαν τα ίδια αποτελέσματα και η έκθεση της Κομισιόν είναι πολύ καλή και δεν θέλουμε σημαντικές παρεκκλήσεις. Η ECR όμως δεν πιστεύει, αντίθετα με τον εισηγητή, ότι εδώ έχουμε το σωστό πλαίσιο για να ρυθμίσουμε σχέσεις δικηγόρου και πελάτη. Αυτό ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο μην είμαστε υπερβολικοί και ρισκάρουμε καθυστερήσεις αν κολλήσουμε στο θέμα αυτό. Επίσης θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να συζητήσουμε για το ύψος των προστήμων. Η Επιτροπή θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο πεδίο εφαρμογής Ε, το συνολικό κύκλο ε, εργασιών. Αυτό είναι το σημαντικό και όχι ο σχετικός κύκλος εργασιών. Διαπιστώσαμε ότι οι επικεφαλής των εθνικών αρχών ε, είπαν ότι έχουν επίσημα αυτονομία αλλά θα πρέπει και τα δημοσιονομικά σχέδια να εγγυώνται και να διασφαλίζουν αυτήν την αυτονομία. Ένα άλλο θέμα σημαντικό για την ομάδα μας οι δημόσιες όπως και οι ιδιωτικές ε, ε, υπηρεσίες θα πρέπει να συμμορφούνται προς τους κανόνες του ανταγωνισμού και να παρακολουθούν την επιρροή που έχει μια επιχείρηση ε, στον ανταγωνισμό. Η ECR ζητεί ανεξάρτητα από το μέγεθος, τα προϊόντα και την οικονομική ισχύ των επιχειρήσεων να ε, γίνεται έλεγχος και να προβλέπονται πρόστιμα. Ε, και αυτό θα ισχύει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ε, αποτρεπτική η ε, ύπαρξη των κυρώσεων. Ε, νομίζω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την Άλντε ο Πιτ Ρίζεκ είναι εδώ, ο Ινωσκιώδη δεν είναι εδώ. Θα μιλήσει κάποιος άλλος για την ομάδα Άλντε. Όχι. Λόμπες Περμέγιο από την Γκουε. Σημεριζόμεθα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό μέσο το οποίο να επιτρέψει στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να παρακολουθούν και να σημειώνουν τις ε, μη σύνομες ενέργειες των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αλλά δεν θα πρέπει όμως ε, να χρησιμοποιείται η πολιτική για την πρόφηση του ανταγωνισμού εις βάρος των εργαζομένων. Οι προτάσεις πάντως είναι χρήσιμες για την καταπολέμηση των καταχρήσεων των ιδιωτικών μονοπωλίων. Θα ήθελα λοιπόν μέσω των τροπολογιών να υπάρξει η δυνατότητα οι αρμόδιες αρχές να αναφέρονται στις εθνικές αρχές ε, για τις δραστηριότητές τους και να μην υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση των δράσεων τους. Πιστεύουμε επίσης ότι η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων προστήμων επί τη βάση ε, του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αλλιώς θεωρούμε ότι οι λογιστικές κομπίνες των πολιεθνικών δεν θα επιτρέψουν παρά την επιβολή ασήμαντων για αυτές ε, ε, πρόστιμα. Θα πρέπει να είναι 2 με 10% τα πρόστιμα αυτά και θα πρέπει να έχουν τα μέσα εφόσον θεωρούν ότι είναι απαραίτητο οι εθνικές αρχές να εισπράττουν τα χρήματα αυτά. Επίσης η αρχή της ευθύνης θα πρέπει να επιβάλλει ε, τα πρόστιμα αυτά να θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγική ε, διαδικασία. Και στα πλαίσια της πρότασης αυτής θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των αρχών επί του ανταγωνισμού για δύο τουλάχιστον χρόνια θα πρέπει να γίνονται δυνατότητες έρευνας για τις σχέσεις ανάμεσα στις αρχές επί του ανταγωνισμού και τις μεγάλες επιχειρήσεις γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις μέσω της διαφθοράς που δημιουργούν είναι γάγκρενα για τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Τα ε, είπα, ακούστηκαν όλα τα επιχειρήματα, αλλά όχι από όλου. Έχει κάνει μια καλή έκθεση ο κύριος Σφάπ. Μπορούμε να συνεργαστούμε λοιπόν επικοδομητικά, μπορούμε να βρούμε για πολλές προτάσεις συμβαστικές λύσεις. Ε, όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι, είμαστε υπέρ της ενίσχυση και διεύρυνση και εδραίωση τη ανεξαρτησία των εθνικών αρχών και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τη δημοσιονομική τους ανεξαρτησία, αλλά και με την επάρκεια του προσωπικού με το οποίο θα επανδρώνονται. Να μην υπάρχει παρέμβαση δηλαδή στις αποφάσεις και για τον προπολογισμό και για την επανδρώση. Θέλουμε επίσης ενίσχυση της διαφάνειας. Πιστεύουμε ότι συμφωνούμε στο στόχο αυτό με τις άλλες ομάδες. Μπορούμε να βρούμε μια λύση. Επίσης για τις αιτήσεις εκθέσεις, για το προσωπικό, για τους πόρους, για τις έρευνες, το αντικείμενο των ερευνών δηλαδή, τη διαφάνεια, υποχρέωση διαφάνεια σε περίπτωση συγκρούσεων συμφερόντων των υπαλλήλων των ερευνητικών αρχών. Θα πρέπει σε όλη την Ευρώπη να ε, υπάρχει διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων ή να αποκαλύπτονται αυτές θα καταθέσουμε μια πολύ σημαντική για μας τροπολογία διάκριση μεταξύ αποζημίωσης και κύρωσης η προστήμου. Αποζημίωση όταν έχει πληγεί στα συμφέροντά του, όταν έχει ζημιωθεί ένας πελάτης, ένας πολίτης. Αυτό δεν μπορεί όμως να αποτελέσει και πρόσχημα για την αποφυγή προστήμου για την παραβίαση του νόμου ούτε αν υπάρχει πρόστιμο να μην υπάρχει αποζημίωση για τους ε, πελάτες. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός δηλαδή και να γραφεί και αυτό στον κανονισμό. Ευχαριστώ. Κυρία Κάπελα από τους ΕΝΦ δεν είναι εδώ, ούτε και κανείς άλλος περισσεύει. Πριν δώσω το λόγο λοιπόν στην Επιτροπή, Καρστιάη, κύριο Σάντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ιδιαίτερα η σημασία έχει και εύστοχη ήταν η έμφαση στη διαφάνεια. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε κάτι άλλο, ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουν και το ρόλο να εξηγούν ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι ένα εργαλείο που ε, ισχύει με, τα ίδια μέτρα και σταθμά πάντα για όλους. Είναι ένας τρόπος εφαρμογής ευρωπαϊκής πολιτικής του ανταγωνισμού για να προσαρμόζεται στις εθνικές πραγματικότητες και αυτό έχει κρίσιμη σημασία για μένα. Το να επιβάλλονται οριζόντια ε, και κεντρικά από βορρά ως νότου και από ανατολής ως δύσεως οι κανόνες του ανταγωνισμού χωρίς περιθώριο για να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές ή περιφερειακές αλήθειες, πραγματικότητες και συνθήκες δεν μπορεί να είναι σωστό. Θα οδηγήσει σε ε, αστάθεια, ανισορροπία, άνισες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν όταν μιλούμε για τις εθνικές αρχές θα πρέπει αυτές να τις βλέπουμε σαν εργαλεία του ευρωπαϊκού δικαίου. Εργαλεία υλοποίησης μιας πολιτικής που θα εφαρμόστε σε όλους αλλά όχι με τρόπο ομοιόμορφο ή ομοιογενή. Απλώς με σκοπό αποτελέσματος. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τους κανόνες διαφάνειας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Επιτροπή, παρακαλώ. Καλό σας απόγευμα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για να πω κάποια πράγματα από πλευράς Κομισιόν. Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί εκτιμούμε και το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΕΚΟΝ που προχώρησε με γρήγορο ρυθμό το φάκελο. Εκτιμούμε όλη την εργασία και την προσεκτική ανάλυση που κάνετε για να ενισχύσουμε την πρόταση που μας απασχόλησε και μας πολύ στην προετοιμασία της και μαζί με τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού. Θα αναφερθώ σε κάποια από τα ζητήματα που θέσατε σήμερα. Καταρχήν, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, να πω ότι βεβαίως συμφωνούμε απόλυτα με την ανάγκη διασφάλισής τους, είναι ζωτικό αυτό, αλλά προσοχή, μην είμαστε πολύ συγκεκριμένοι όταν μιλούμε για την επαφή δικηγόρου-πελάτη, ε, και γιατί αυτά είναι, υπάρχουν στα εθνικά συστήματα. Ε, ε, αναφέρονται σε άλλους τομείς εκτός από τον ανταγωνισμό και ρυθμίζονται διαφορετικά από τα κράτη-μέλη. Εδώ χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Τώρα, η σημασία των ε, περιστρεφόμενων θυρών, όταν περάσουμε δηλαδή από την αρχή ανταγωνισμού σε μια ε, δικηγορική εταιρεία, είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και κάποιος που φεύγει από την ε, αρχή ανταγωνισμού δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στις υποθέσεις τις ίδιες ε, όπως και πριν. Συμφωνούμε εδώ, αλλά και εδώ χρειάζεται προσοχή. Δεν πρέπει να είμαστε πολύ υπερβολικά συγκεκριμένοι. Σίγουρα δεν υπάρχει μία λύση που να ισχύει παντού. Ε, υπάρχει κίνδυνος όταν μπαίνουμε σε μεγάλες λεπτομέρειες ε, ε, αντιμετώπιση σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή ποιο είναι, ποιο είναι το εύλογο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν μπορεί κανείς να απασχοληθεί στην ίδια υπόθεση ε, ως δικηγόρος όπως όταν ήταν στην αρχή ανταγωνισμού. Ε, πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία και αυτό αναφέρθηκε σήμερα. Υπογραμμίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις. Η πρόσβαση είναι πολύ σημαντική λέξη γιατί πρόκειται για αποθήκευση στον νέφος. Στην ψηφιακή εποχή θα πρέπει οι αρχές ανταγωνισμού να μπορούν να ε, επιβάλλουν τις αποφάσεις και γι' αυτό να βρίσκουν τις ε, πληροφορίες για τις παραβιάσεις. Τέλος, για το μέγιστο πρόστιμο και το σχετικό κύκλο εργασιών, να πω ότι όταν πρόκειται για τα πρόστιμα, ο στόχος μας ήταν να απαλείψουμε οποιαδήποτε εμπόδια που υπάρχουν στα εθνικά δικαιικά συστήματα και που εμποδίζουν τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού από την επιβολή αποτρεπτικών προστήμων ο στόχος αυτής της πρότασης δεν είναι η εναρμόνιση, αλλά η απάλληψη των εμποδίων. Γι' αυτό θεωρούμε, ή μάλλον γι' αυτό δεν θεωρήσαμε κατάλληλο να εναρμονίσουμε το μέγιστο ποσό των προστήμων. Θέλαμε τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να προχωρήσουν περισσότερο. Γι' αυτό άλλωστε θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι όταν υπολογίζουμε το το ποσό, τουλάχιστον 10%, η Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού μπορεί να λάβει υπόψη το συνολικό κύκλο εργασιών, γιατί όπως είπατε και εσείς, αυτό είναι το σημείο αναφοράς για την οικονομική ισχύ των εταιριών και αυτό χρειάζονται οι αρχές ανταγωνισμού για να μπορούν να επιβάλλουν αποτρεπτικά πρόστιμα. Σταματώ εδώ και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ δεν ε, υπάρχει κάτι άλλο. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και τη συζήτηση. Ε, η ψηφοφορία θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Διακοπή 15 λεπτών. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου της κυρίας Μπερές. Ε, μπορείτε να επαναλάβετε ο χρόνος για τη συζήτηση ήταν σαφής. Αν είσαστε ε, από την αρχή ήταν δύο λεπτά οι ερωτήσεις, τρία λεπτά οι απαντήσεις και όλοι θεώρησαν ότι θα τελειώνει στις τέσσερις. Θα μπορούσατε να είσαστε εδώ από την αρχή. Μα δεν έφυγα. Ήμουν εδώ συνέχεια. Παραπονούμε για την ακρόαση ΠΕΠ, γιατί ε, θα μπορούσε να γίνει περισσότερη συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες. Δεν μπορούσα να παρέμβω και να αναλύσω περισσότερο τα θέματα γιατί μας είπατε ότι δεν προλαβαίναμε και τώρα κάνουμε διάλειμμα. Αυτή την παρατήρηση ήθελα να κάνω ότι δεν μου δόθη ο λόγος ενώ τώρα διακόπτουμε. Όποιο ε, ε, λοιπόν, τώρα ε, θα κάνουμε μια διακοπή για 15 λεπτά. Ευχαριστώ.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

So, uh, Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Θέλω να καλωσορίσω την ε, Μάργαρετ Βέστραγκερ την αρμόδια επίτροπο για θέματα ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα στο δεύτερο διαφθρωτικό διάλογο του 2017. Η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο θα μας δώσει την ευκαιρία να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις ε, στα θέματα των δραστηριοτήτων και των ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στα θέματα που έχουν σχέση με τις τράπεζες και την ψηφιακή οικονομία. Είναι σημαντικά θέματα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας μέχρι τώρα και για τις δραστηριότητές σας ε, ε, σας δίνουμε αμέσω το λόγο. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε ξανά. Σας ευχαριστώ για την θερμή σας υποδοχή. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Ραμόν Τρεμόσα και τους Σκιώδης για την υποστήριξή τους στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού είναι θετικό να βλέπει κανείς ότι συμφωνούμε ότι η πολιτική επί του ανταγωνισμού είναι κάτι το οποίο λειτουργεί. Ε, μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες ε, κρατώντας ανοιχτές τις αγορές και οι πολίτες ε, να βλέπουν ακριβώς την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων από πλευράς των επιχειρήσεων με διαφάνεια και με δυνατότητες επιλογής. Αυτό το οποίο βρίσκω εγώ σαν κάτι θετικό είναι ότι πράγματι πρέπει να ληφθούν μέτρα αυστηρά κατά των παραβιάσεων του ανταγωνισμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα δώσει στους πολίτες την εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία επιθυμούμε. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς οι οποίοι ελπίζω να σας ενδιαφέρουν. Θα αναφερθώ στην περίπτωση του Google, θα μιλήσουμε για τα φάρμακα, θα μιλήσουμε για τις τράπεζες, θα μιλήσουμε για τους φόρους και για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Ειδικά για την Google, εμείς τον μήνα Ιούλιο πήραμε την πρώτη απόφαση αντιτράστ εναντίον της Google, και κυρίως του Google Shopping. Αυτό το οποίο βρήκαμε είναι ότι το Google Search συστηματικά ευνοούσε τα αποτελέσματα Google Shopping σε σχέση με τις υπόλοιπες ε, υπηρεσίες αγορών διαδικτυακά. Αυτή είναι μια κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης ε, της Google και επιβάλαμε ένα πρόστιμο 2,4 δις ευρώ. Τώρα η Google θα πρέπει να δώσει εγγυήσει ότι το Google Shopping θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως οι ανταγωνιστές. Η Google προτείνει λύσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου. Παρακολουθούμε τις ε, ε, προτάσεις αυτές. Έχουμε τεχνικούς εμπειρογνώμονες ε, μετά από διαγωνισμό προέρχονται από την επιχείρηση Mavens και θα τους χρησιμοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε για να υπάρχει σωστή συνεργασία. Βέβαια αυτό δεν κλείνει την υπόθεση. Εμείς συνεχίζουμε τα επιχειρήματά μας σε σχέση με την χρήση του Android ε, στα πλαίσια της πλατφόρμας AdSense που χρησιμοποιεί η Google για να πωλεί ε, διαφημίσεις. Είναι υποθέσεις οι οποίες για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα. Απαιτείται οι αγορές να είναι ανοιχτές, να λειτουργούν ισότιμα και όχι μόνο στην ψηφιακή οικονομία, αλλά για όλες τις ε, επιχειρήσεις και online και offline. Όταν ένας πολίτης αρρωσταίνει και χρειάζεται φάρμακα, θα μπορεί να παίρνει τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται. Ε, αυτό λοιπόν είναι έχει σχέση με την αγορά η οποία είναι παλαιού τύπου αλλά είναι ταυτόχρονα και πολύ περίπλοκη και μεγάλου μεγέθους. Εμείς ξεκινήσαμε λοιπόν την δράση μας για κατάχρηση κυρίαρχης θέσης από τη φαρμακευτική επιχείρηση Aspen σε σχέση με πέντε φάρμακα για την καταπολέμηση του καρκίνου δυστυχώς επέβαλε μερικές φορές αυξήσεις για τα προϊόντα αυτά εκατοντάδες, ε, γενικά τεράστιες αυξήσεις, 100% πιο ακριβά. Οι αυξήσεις στην Ιταλία σαν παράδειγμα σε σχέση με τις τιμές της Άσπεν ήταν υπερβολικές και αδικαιολόγητες. Είναι η πρώτη περίπτωση που έχουμε εμείς για υπερβολικές τιμές στη φαρμακευτική βιομηχανία και θα επενδύσουμε στο θέμα αυτό ερευνητικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και για μας. Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις επενδύσεις, στην καινοτομία και στην δυνατότητα απόσβεσης της συγκεκριμένης επένδυσης. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα και με συγκεκριμένους όρους. Ε, επίσης μας απασχόλησαν και τα θέματα των πιστοτικών ιδρυμάτων. Ελήφθησαν ορισμένες αποφάσεις. Έτσι και αλλιώ είναι υποχρέωσή μας να εξετάζουμε την κατάσταση των μεμονωμένων τραπεζών και ο νομοθέτης αυτό το οποίο προβλέπει είναι κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες. Αν μία τράπεζα δεν είναι βιώσιμη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο εποπτικός μηχανισμός χαρακτηρίζουν την τράπεζα αυτή ε, σαν τράπεζα η οποία θα προχωρήσει σε διαδικασίες πτώχευσης ή εξυγίανσης και ε, ο, ο μηχανισμός αν θέλετε ο οποίος υπάρχει, ο ενίος μηχανισμός θα κρίνει τον τρόπο με τον οποίο θα εξηγιανθούν οι συγκεκριμένες τράπεζες. Αυτό σημαίνει, συνέβη και με τις δύο τράπεζες Βένετο σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ε, πτώχευσης. Εμείς εγκρίναμε την βοήθεια για να περιορίσουμε ε, το, τις συνέπειες το, της αλλαγής της κατάστασης της τράπεζας αυτές στην περιφερειακή οικονομία έγινε το λεγόμενο bail-in για να μειωθεί άλλωστε και η κρατική βοήθεια η οποία θα χρειαζόταν. Είναι βασικό ότι οι τράπεζες θα πρέπει να δημιουργήσουν αρκετά προστατευτικά μέσα για να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες και να αποφεύγουν την ανάγκη κρατικής βοήθειας. Ένα από τα θέματα τα οποία επηρεάζουν το εάν οι πολίτες μας μας εμπιστεύονται και εμπιστεύονται την οικονομία μας έχει σχέση με την φορολογία. Τα τελευταία στοιχεία είναι τα λεγόμενα Paradise Papers. Αυτά τα Paradise Papers περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τις φορολογικές ρυθμίσεις πολλών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως και με τα προηγούμενα Panama Leaks, οι υπηρεσίες μας εξετάζουν τις πληροφορίες αυτές πάρα πολύ προσεκτικά. Αν βρούμε λόγους οι οποίοι θα μας ανησυχήσουν, θα ξεκινήσουμε περισσότερες έρευνες επί τη βάση των πληροφοριών αυτών. Ε, εμείς εξακολουθούμε νομίζω με την δράση μας να παράγουμε αποτελέσματα. Τον προηγούμενο μήνα διατάξαμε το Λουξεμβούργο να ανακτήσει 250 εκατομμύρια ευρώ απλήρωτους φόρους από την Amazon. Δυστυχώς θα έπρεπε, να παραπέμψουμε την Ιρλανδία στο δικαστήριο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάκτησης φορολογικών εσόδων από την εταιρεία Apple. Ε, υπήρξε ανάκτηση φόρων σε άλλες ε, περιπτώσεις ε, όπως και στο Βέλγιο και σε άλλες 35 περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτές είναι οι περιπτώσεις με τις οποίες ασχοληθήκαμε. Υπάρχουν και νέες περιπτώσεις που μας απασχολούν. Δύο εβδομάδες ξεκινήσαμε διαδικασίες κρατικής βοήθειας εις βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου οι κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου για εταιρείε που ελέγχονται από το εξωτερικό έχουν σαν στόχο την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Αυτό δεν είναι κακό. Αλλά από ό,τι φαίνεται ε, και αυτό που μας ανασυχεί είναι ότι στην ουσία αντιμετωπίζουν ορισμένες επιχειρήσεις με προτιμησιακό τρόπο. Ε, δηλαδή υπάρχουν μέτρα που δεν ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι έχουμε μπροστά μας αρκετές δυσκολίες οι διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα και φυσικά αυτό δεν είναι μόνο θέμα κρατικών επιδοτήσεων, απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες να καλύπτουν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την καθοδήγηση του Πιεύ Μοσκοβισή. Κάποια από τα θέματα με τα οποία ασχολούμεθα και στα οποία προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις είναι το πώς η παγκοσμιοποίηση ουσιαστικά θα δουλέψει για μας. Υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν δυνατότητες και κάποιες από τις πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνουμε και παίρνουμε και από κοινού έχουν σαν βασικό στόχο την αναδιανομή αν θέλετε των ευκαιριών που παρέχει η παγκοσμιοποίηση. Δεν είναι δεδομένο ότι η παγκοσμιοποίηση εξυπηρετεί όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο. Αν δεν ελέγξει κανείς ε, τους, ε, τα θέματα της ε, παγκοσμιοποίησης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ορισμένους πολίτες ευνοώντας ίσως κάποιους άλλους. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε αυτούς τους τομείς θα πρέπει να καταστήσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ικανές να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ότι έχουμε αυτά τα οποία χρειάζεται η Ευρώπη. Έχουμε έξυπνα μυαλά, έχουμε δυνατότητες, έχουμε πολύ καλή έρευνα και ιδιωτική και δημόσια. Έχουμε ένα περιβάλλον επιχειρηματικό αξιόπιστο, προβλέψιμο και γι' αυτό η Ευρώπη θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά με σωστό τρόπο, να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, να ανοίξει νέες ευκαιρίες έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει να ευημερήσει. Εμείς δεν θέλουμε να ευνοήσουμε ορισμένες επιχειρήσεις εις βάρος άλλων. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε τις σωστές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες. Γι' αυτό θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την θέση των πολιτών μας έτσι ώστε να μην φοβούνται την παγκοσμιοποίηση. Και εδώ οι κανόνες του ανταγωνισμού παίζουν κάποιο ρόλο. Ο ανταγωνισμός και οι κανόνες για τον ανταγωνισμό ενισχύουν τους πολίτες. Αν αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αν δεν κάνουν αυτά τα οποία θέλουν οι πολίτες, οι πελάτες θα πάνε κάπου αλλού σημαίνει ότι, δεν σημαίνει μάλλον ότι θα πρέπει να αποκεντρώσουμε ε, την επιβολή ε, του ανταγωνισμού, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το τι ισχύει σε όλους τους τομείς. Τώρα, για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων. Ε, οι συγχωνεύσεις και ο έλεγχος των συγχωνεύσεων δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαγορεύσουμε στις επιχειρήσεις να είναι μεγάλες. Μπορεί κανείς να είναι μεγάλος και να είναι επιτυχής στην Ευρώπη. Το μέγεθος μπορεί να είναι και κάτι καλό για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Όταν έχεις επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιο καινοτόμες, έχουν περισσότερους πόρους, περισσότερες δυνατότητες, γίνονται και πιο ελκυστικές για τους πελάτες τους. Το θέμα είναι ότι όταν βλέπουμε το σύστημα πώς λειτουργεί, βλέπουμε ότι όταν ότι ε, όταν έχουμε περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων οι αγορές να εξυπηρετούν το σύνολο των ε, εμπλεκομένων και όχι μόνο τις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις. Η παγκοσμιοποίηση εδώ ε, είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τα πάντα ότι κάνουμε. Το 60% των περιπτώσεων συγχωνεύσεων που αντιμετωπίζουμε έχουν να κάνουν εν με την παγκοσμιοποίηση και το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Το θέμα δεν είναι βέβαια το τι συμβαίνει γενικά, το ποιε είναι οι τάσει. Το θέμα είναι τι συμβαίνει κατά περίπτωση. Σε πάρα πολλά θέματα, σε επιμέρους, σε, στις μεταφορές, στα τρόφιμα, στον καφέ, στα πάντα. έτσι ώστε οι αγορές να εξυπηρετούν τους πολίτες. Εμείς δεν προστατεύουμε τις επιχειρήσεις, προστατεύουμε τους πολίτες. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά της κάθε δραστηριότητας. Το τσιμέντο είναι πάρα πολύ ακριβώς στις μεταφορές και δεν έχει νόημα πολλές φορές να συγκρίνει κανείς το σκυρόδεμα το οποίο παράγεται από πάρα πολύ μακριά, γιατί αν παράγεται πάρα πολύ μακριά, ώσπου να έρθει στην Ευρώπη θα γίνει πάρα πολύ ακριβό, οπότε πάρα πολύ απλά δεν έρχεται. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουμε την κάθε αγορά με ξεχωριστό τρόπο. Τα τελευταία δέκα χρόνια λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει πάνω από 3.000 συγχωνεύσεις, έχει μπλοκάρει μόνον 7 συγχωνεύσεις. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι στις, περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται κάποιες λύσεις επιτρέποντας τις συγχωνεύσεις να προχωρήσουν, προστατεύοντας τον ανταγωνισμό στην αγορά ταυτόχρονα. Και πολλές ε, από τις συγχωνεύσεις αυτές έχουν αδειοδοτηθεί λοιπόν και οδήγησαν στην δημιουργία Ευρωπαίων πρωταθλητών σαν παράδειγμα Γκαμέζα και Siemens στον τομέα των αιωλικών τουρμπινών. Νομίζω ότι έχουμε και σε άλλους τομείς όπως στα τρόφιμα πολύ μεγάλες επιτυχείς ευρωπαϊκές εταιρείες. Danone και White Wave. Ε, βλέπετε λοιπόν πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορεί να επηρεάζουν και την παγκοσμιοποίηση από μόνες τους. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε διπλό στόχο. Πρώτον, επιτυχείς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια σκηνή και ταυτόχρονα να υπάρχει ανταγωνισμός στην Ευρώπη, ανοιχτές αγορές για όλους και ίσες ευκαιρίες ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, αυτό το κάνουμε συνεργαζόμενοι με τις εθνικές επί του ανταγωνισμού αρχές και γι' αυτό ακριβώς στο τέλος της παρέμβασής μου θέλω να σας συγχαρώ, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόοδο που έχετε σημειώσει στην πρόταση ECN+. Νομίζω ότι κάνετε μια εξαιρετική δουλειά για τους πολίτες και για τα κράτη-μέλη. Είμαι ευγνώμων για τη συμμετοχή σας στις προσπάθειές μας και επίσης ε, και για τον σεβασμό που δείχνεται απέναντι στις αρχές επί του ανταγωνισμού. Γιατί αλλιώς ε, η επιβολή του νόμου σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα ήταν εφικτή. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα και για σας και νομίζω ότι όταν εφαρμόζεται το δίκαιο επί του ανταγωνισμού εξυπηρετούνται οι πολίτες. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής μας εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιακό ο κατάλογο των δραστηριοτήτων σα. Και βεβαίως είναι ουσιώδες στοιχείο της ενιαία αγοράς, η πολιτική του ανταγωνισμού. Ιδιαίτερα τώρα και με τις διαπραγματεύσει για τον Brexit δεν είναι δυνατόν να αποκοπεί από την ε, πολιτική ανταγωνισμού ενιαία αγορά. Όπως είπατε και εσείς, μια καλή πολιτική ανταγωνισμού μπορεί και να ενισχύσει τη θέση του πολίτη και να τον συμφιλιώσει με την παγκοσμιοποίηση και αφετέρου να διαμορφώσει, να συνδιαμορφώσει την παγκοσμιοποίηση. Φορολόγηση, συγχωνεύσεις και ούτω καθεξής. Πρόκειται για ένα κέριο τομέα, ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ισχυρό. Όχι ε, επαρκές, αλλά πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην καλή πολιτική ανταγωνισμού. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να υποστηρίζουμε τη πολιτική που ακολουθείτε μέχρι τώρα και συνεχίζουμε και εμείς την προσπάθειά μας στα πλαίσια της πρότασης CCN+. Συζητάμε τις διάφορες τροπολογίες και νομίζω ότι θα περάσουμε στην τελική ψηφοφορία μας τον μήνα Φεβρουάριο. Λοιπόν συνάδελφοι ξεκινάμε τις παρεμβάσεις. Ο Φέρμπερ της Ομάδας για τον Ανταγωνισμό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Δίκαιο του Ανταγωνισμού Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την καλή ε, συνεργασία. Ο Γενικός σας Διευθυντής είχε έρθει πριν από δύο εβδομάδες για πολύ εντατική ανταλλαγή ε, απόψεων και γενικά έχουμε πολλές επαφές ε, και καλές επαφές. Δύο σημεία θα θίξω. Ο ΣΑΣ, ένα έγγραφο εργασίας πρόσφατα για το αλγόριθμι και συμπράξεις, algorithms and collusions, έθεσε ένα θέμα σε σχέση με την επιρροή των αλγορίθμων. Πολλές επιχειρήσεις επενδύουν στους αλγορίθμους για δυναμική, δυναμικό καθορισμό τιμών, ε, διότι υπάρχει ανάγκη προσαρμογής στις ανάγκες. Ε, ε, επηρεάζει η πολιτική ανταγωνισμού τον καθορισμό της βέλτιστης τιμής. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα και στη Γερμανία. Ένας ανταγωνιστής έφυγε από την αγορά και μπορούμε να δούμε πώς ε, έγινε αυτό. Ε, όταν δύο ή περισσότεροι αλγόριθμοι αλληλεπιδρούν, ε, ο καθορισμός της τιμής δεν λαμβάνει υπόψη τον καταναλωτή και αν υπάρχουν και συνεννοήσεις και συμπράξεις για τις τιμές δημιουργείται καρτέλ. Μιλήσατε και για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων, ένα θέμα που πάντα μας ενδιέφερε πολύ. Θυμίζω τη συγχώνευση Facebook και WhatsApp, το θέμα της αξιολόγησης των δεδομένων επίσης. Το προηγούμενο έτος και μέχρι τον Ιανουάριο τον, επόμενο, ε, από τον προηγούμενο χρόνο και μέχρι τον Ιανουάριο φέτος κάνατε πολλές διαβουλεύσεις για την αξιολόγηση των ε, δεδομένων και, κάνατε, ε, και δεν ξέρω εάν μπορείτε να μας πείτε εάν καταλήξατε σε κάποια συμπεράσματα σχετικά. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και εγώ διότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συνεργασία μας που μας προχωρεί και μας βοηθεί στη δουλειά μας. Θέλουμε να ξέρουμε τις γνώμες σας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή εποχή για να συζητήσουμε σε βάθος πώς βλέπουμε τις τεχνολογίες αυτομάθησης και τους αλγόριθμους και τι ρόλο παίζουν. Ε, θα πρέπει βέβαια οι αλγόριθμοι να μελετηθούν πολύ, διότι θα πρέπει να μας επιτρέπουν να δούμε τι θα κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είδα ένα πείραμα, ε, ήταν μια εικονική, ε, ένα, ε, μια, στίβος για πάλι με δύο ρομπότ που δεν μπορούσαν να περπατήσουν στην αρχή, να κινηθούν, μετά από δισεκατομμύρια δοκιμές και σφάλματα, αυτά τα εικονικά ρομπότ έμαθαν όχι μόνο να ε, κινούνται, αλλά και την πάλι όλη την τακτική, τα χτυπήματα κλπ. Ενώ άρχισαν από το μηδέν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του τι μας περιμένει όταν έχουμε τεχνολογίες μάθησης στη διάθεσή μας. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι όχι ε, ο αλγόριθμος ε, ε, ε, έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Εσείς είστε υπεύθυνο για τον αλγόριθμο και τα αποτελέσματα. Πρέπει να ξέρετε τα υπέρ και τα κατά τις οδηγίες και τους περιορισμούς που θα δώσετε στον αλγόριθμο για ε, το δυναμικό καθορισμό τιμών και για την εποπτεία των αγορών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της παλιάς σχολής η οποία ε, εξέταζε ας πούμε τον ε, κάποιο σταθμό καυσίμων και πώς καθορίζει τις τιμές και τι... Ε, διαφοροποιεί τις τιμές από τον ένα σταθμό στον άλλον. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τον ανταγωνισμό όπως διαμορφώνεται στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε τώρα τη μελέτη όλων αυτών. Γι' αυτό άλλωστε και ο ΩΣΑ ασχολείται με το θέμα. Τώρα για τα δεδομένα εμείς ετοιμαζόμαστε για την πρώτη υπόθεση μεγάλων δεδομένων, εξετάζοντας ζητήματα δεδομένων σε κάποιες από τις υποθέσεις μας. Και ευτυχώς το κάναμε αυτό, γιατί κάναμε ανάλυση στο Facebook και τι θα γίνει αν συνδυαστούν τα δεδομένα. Αν και έλεγαν ότι κάτι τέτοιο δεν θα, συμβεί. Κάναμε ανάλυση και είδαμε ότι δεν θα ήταν φραγμός για την είσοδο άλλων στην αγορά αυτή. Ε, αυτό είναι ένα ζήτημα ουσίας. Τα δεδομένα που έχει μια εταιρεία, αν γίνονται εμπόδια για την είσοδο στην αγορά άλλων, αυτό είναι θέμα. Ε, νομίζω ότι το ε, πιο προφανές παράδειγμα είναι ένα γαλλικό που οι γαλλικές αρχές ανταγωνισμού ε, ε, είπαν ότι ένας ε, πάροχος ενέργειας θα έπρεπε να μοιραστεί δεδομένα, διότι είχαν βάση πελατών και η μη, της η, η μη κοινοποίηση της βάσης των πελατών δημιουργεί εμπόδιο στην αγορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και για την καινοτομία. θα πρέπει να μην υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο. Αυτό μπορούμε να το δούμε ε, αυτό είναι σίγουρα ε, ένα πράγμα για το οποίο ετοιμαζόμαστε. Αλφρεντ Σαντ. Οι κανόνες για τις κριτικές επιδοτήσεις στόχο έχουν να αποτρέψουν τον ε, θέμα τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο βλέπουμε ότι είναι άνησες οι συνθήκες στην παγκοσμιοποιημένη αγορά με κρατικές επιδοτήσεις, ρυθμιστικές ε, παρεμβάσεις και στον εργασιακό χώρο αλλά και στον περιβαλλοντικό. Τέτοιες διαφορές λοιπόν είναι ορατές και στο σενάριο των ε, αεροπορικών εταιριών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Lufthansa, παραδείγματι, ισχυρίζεται ότι έχει χάσει τον τρίτο η Lufthansa από την αγορά εργασίας της από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη από το 2005 τι συμβαίνει στην ε, περιοχή, στον τομέα αυτών και τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε. Βλέπετε κάποια λύση και τι είδου μορφή μπορεί να πάρει αυτή. Και πάλι σε αεροπορικέ μεταφορέ. Ε, ενημερωθήκαμε τον προηγούμενο μήνα ότι είχε εξαγοράσει την Air Berlin η Lufthansa ύστερα από την πτώχευση της ε, τον προηγούμενο Αύγουστο. Εν τω μεταξύ όμως τη Ryanair ισχυρίζεται ότι πρόκειται για μια συνωμοτική εξαγορά για να ενισχυθεί ο εθνικός αερομεταφορέας. Άλλοι ισχυρίζονται ότι ενισχύεται η ε, θέση στην αγορά της ε, Lufthansa και της, ε, του ομίλου Star Alliance. Έχει Επιτροπή κάποια γνώμη γι' αυτό και για τη συγχώνευση. This is uh, this is a very important market, not only... Ναι, είναι πολύ σημαντική αγορά, όχι μόνο για το κλάδο, αλλά για τον πολίτη. η επανάσταση με τις αερομεταφοράς τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει, τις έχει αλλάξει την κατάσταση για πάρα πολλούς πολίτες. Έχουν μειωθεί οι τιμές, επιτρέπουν έτσι να ταξιδεύουν όλο και περισσότεροι πολίτες. Όταν εγώ ήμουν μικρή πηγαίναμε με το αυτοκίνητο στο Χάτσον. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά μου σήμερα και λυπούμε ε, Μάρκο που το λέω αυτό. Αν έπρεπε να κάνουμε τόσε ώρε δρόμο με το αυτοκίνητα. παιδιά μου θα αισθανόταν πολύ μεγάλη απογοήτευση. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία και ρόλο. Βέβαια στη δική μα τη δουλειά ο τομέα των αερομεταφορών. Η συνάδελφο ε, Βιολέτα Μπούρτ ε, ιδιαίτερα ασχολείται με τα θέματα των αερομεταφορέων από τον Περσικό κόλπο και του Ευρωπαίου Αερομεταφορέ για να εξασφαλίσει θεμητέ συνθήκε ανταγωνισμού γιατί πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχουν κάποιε ανησυχίε και μελήματα για συνθήκε ανταγωνισμού από ε, τρίτου αερομεταφορείς, τρίτων χωρών δηλαδή. Ε, υπάρχει λοιπόν εντολή για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ, όπου εδρεύουν μεγάλοι αεροπορικοί αερομεταφορής ε, για συμφωνίες που θα μας επιτρέψουν περισσότερη διαφάνεια, τη μέγιστη δυνατή που είναι απαραίτητη. Στο δικό μας βέβαια ε, το θεματολόγιο παρακολουθούμε ιδιαίτερα τις συμφωνίες παροχής αερομεταφορών ή υπηρεσιών αερομεταφορών, εάν είναι θεμητός ανταγωνισμός, στον χώρο των συγχωνεύσεων Παρακολουθούμε βέβαια και τι συγχωνεύσει μεταξύ αεροπορικών ε, εταιριών. Για τη συγχώνευση Lufthansa και Air Berlin τώρα, Πρόκειται για μια αγορά που εξετάζουμε πολύ μεγάλη προσοχή και διαπιστώνουμε κάποιες πολύ σοβαρές συμπτώσεις. Ε, στο ιστορικό της Γερμανίας, σε παραδείγμα, τη διαγνώσκεται κίνδυνος ε, στρέβλος του ανταγωνισμού σε, πολλούς, σε πολλά δρομολόγια, σε πάρα πολλά δρομολόγια, άρα μπορεί να οδηγηθούμε σε χαμηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και υψηλότερες τιμές. Ήδη από το γεγονός και μόνο ότι η Air Berlin δεν δραστηριοποιείται στην αγορά πλέον, το ότι είναι στο έδαφος τα αεροπλάνα της, επηρεάζει και τους μηχανισμούς σχηματισμού τιμών. Εμείς είμαστε επιτροπές, επιτροπή δεν ορίζουμε τιμές, εννοείται ότι, ότι οι επιχειρήσεις ορίζουν τις τιμές τους. Αλλά βλέπουμε αμέσως ότι αντέδρασαν οι αγορές όταν δεν εξυπηρετούνται πλέον κάποια δρομολόγια και μένουν στο έδαφος τα αεροπλάνα. Για να μπορέσουν λοιπόν να συνεχιστούν στο δυνατόν περισσότερα αεροπορικά δρομολόγια, κάναμε μια αρχική εξαίρεση, παρέκκληση από τις διαδικασίες μας για να αποτρέψουμε τον κίνδυνο του ε, αυτόματου dumping με την έννοια ότι ορισμένα αεροπλάνα της Air Berlin ήδη είχαν μπει σε δρομολόγια της Lufthansa. Για να μην σταματήσουν λοιπόν αυτά τα δρομολόγια, ε, επιτρέψαμε να συνεχιστούν υπό τη σημαία της Λουσχάνης, αλλά ταυτόχρονα παρακολουθούμε τις εξελίξεις για να δούμε τι συμβαίνει αν, σε μια συγχώνευση, αν από μια συγχώνευση προκύψει ε, απουσία ανταγωνισμού για ορισμένα δρομολόγια. Αυτό κάνουμε τώρα με πολύ αυστηρές προδιαγραφές και προθεσμία συγκεκριμένα. Για να δούμε ποια είναι η κατάσταση και πώς διαμορφώνει η αγορά για τον ε, καταναλωτή έχουμε προβλέψει αρχές Δεκεμβρίου να ε, εξετάσουμε πώς έχει προχωρήσει η κατάσταση. Ευχαριστώ κυρία Σουίνμπερν. Πρόεδρε, ευχαριστώ και κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι εκφράζω τους συναδέλφους λέγοντας ότι είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονε για αυτόν τον διάλογο και τις ουσιαστικέ απαντήσεις που μας δίνετε που δεν ε, παίρνουμε πάντα από όλους τους επιτρόπους. Θα ήθελα τώρα να εκθέσω ένα θέμα λεπτό που συστήσαμε και χθε με τον πρόεδρο Ντράγκη, το έθεσε ένα συνάδελφος, για τις δράσεις που πρόσφατα έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με το πρόγραμμα εξαγοράς ομολόγων ε, των εταιριών, το CSPP, όπως ε, το, είναι το ακρονίμιο του, επιτρέπει την εξαγορά ε, ομολόγων που δεν έχουν εκδώσει τράπεζες από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ. 92 δις ευρώ συνολικά, 11% των διαθέσιμων και επιλέξιμων ομολόγων. Αυτό όμως μπορεί να έχει ε, επίδραση στον ανταγωνισμό και σε άλλους που θα ήθελαν ενδεχομένω να αγοράσουν αυτά τα ομολόγα που έτσι βγαίνουν έξω από την αγορά και αυτό επηρεάζει γενικά την αγορά ομολόγων. Από τις ε, απαντήσεις σε ερωτήσεις άλλων συναδέλφων ε, από τον Μάριο Ντράγκη είδαμε ότι αυτό το σύστημα, αυτό το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ε, απέβει προς όφελος μάλλον μεγάλων επιχειρήσεων και όχι των μικρομεσαίων. Και έτσι, δεδομένου ότι αποκλείονται από τις διατάξεις για κατάχρηση δεσπόσου θέσης ή αγοράς οι δράσεις της ΕΚΤ, ε, μήπως εξετάζονται τουλάχιστον υπό το πρίσμα του δικαίου του ανταγωνισμού. Και όταν υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει μια επιλογή να κάνει πολύ σημαντική σε σχέση όμως και, τη, με την ε, αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων. Αυτό κάνει η ΕΚΤΑ ή, ή αγοράζει ομόλογα γενικά οριζόντια, δηλαδή κατά ποσοστό ανάλογα του κράτους ή της επιχείρησης. Απάντηση. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν έχω απάντηση για την ερώτησή σας η ΕΚΤ δεν μπορεί να θεωρηθεί επιχείρηση υπό την έννοια του δικαίου μας. Είναι ένα σουιγκέρερης πλάσμα, για να το πω έτσι. Και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει ευθέως στο πεδίο δραστηριοτήτων μας. Επομένως, δεν ξέρω ποια θα ήταν μια καλή απάντηση Αντιλαμβάνομαι εσείς που το πάτε και πώς βλέπετε τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω τι προσέγγιση δικαίου του ανταγωνισμού θα μπορούσε να έχει κανείς έναντι ενός προγράμματος αγοράς ομολόγων και με ποια βάση. Ούτε καν τι κατευθυντήριες γραμμές ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όταν επιλέγει ποια θα αγοράσει ή ποια δεν θα αγοράσει αλλά θα το μελετήσω και θα επανέλθω με κάτι πιο συγκεκριμένο ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε βέβαια για ε, εταιρικά ομόλογα, επενδυτικά Οπότε είναι μια ειδικού τύπου χρηματοδότηση. Και δεν ξέρω τι επίπτωση έχει αυτό στον ανταγωνισμό. Αλλά θα περιμένουμε απάντηση στο ερώτημα αυτό. Κύριε Στρεμόζο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γουαλτιέρη και καλησπέρα. Καλησπέρα σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν ε, συμφωνώ μαζί σας σε σχέση με Apple και Amazon στο Λουξεμβούργο. Είναι θέμα φορολογικής δικαιοσύνης και κάνετε πολύ καλή δουλειά εκεί όπως και αλλού. Ε, η Kate Swinburne έκανε τη μία μου ερώτηση για το πρόγραμμα αγορών. Ήθελα να σας ρωτήσω επίσης σε σε αυτά τα πλαίσια, γιατί θα δείτε ότι πολλά μέλη της Επιτροπής μας ανησυχούν σχετικά με τον ανταγωνισμό στις μεταφορές. 44 βουλευτές αυτής της Επιτροπής, μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή, έστειλε επιστολή πέρσι τον Ιούνιο, ζητώντας διαφάνεια από την ΕΚΤ. Θέλαμε να ξέρουμε ποιες ε, κεντρικές τράπεζες ε, αγόραζαν ε, τι από τις εταιρείε. Και μετά πήραμε έναν κατάλογο, αφού έγραψε και ο τύπος. Ξέρω ότι τον κατάλογο τον έχετε από τον Ιούλιο και ανακαλύψαμε για παράδειγμα ότι η Ιρλανδία, η κεντρική τράπεζα δηλαδή εκεί, αγόραζε ε, χρέος της ε, Ryanair. Δεν θα επισέλθω στις λεπτομέρειες της σκοπιμότητας αυτών των αγορών, αλλά νομίζω ότι έτσι διαστρεβλώνονται οι ίσοι κανόνες του ανταγωνισμού. Γιατί, εμείς επικρίνεται, γιατί επικρίνεται η Ιταλία, για παράδειγμα, που βοηθάει την Αλιτάλια με κρατικές ενισχύσεις. Αλλά η Banco Italia... δεν αγόρασε ε, μέρος του χρέους της Αλιτάλια. Έτσι λοιπόν η ΕΚΤ δημιουργεί στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτή τη γνώμη έχουμε αρκετοί από εμάς. Μπορούμε να πούμε δηλαδή στην έκθεση ότι δεν συμφωνούμε με αυτά που συμβαίνουν με την Ερμπερλίν, τη Λουφτχάνσα και την Ελιτάλια, αλλά από την άλλη έχουμε το πρόβλημα αυτό. Οι υπηρεσίες σας λοιπόν παρακαλώ θα έπρεπε να μελετήσουν το ζήτημα διότι θα ε, αναλάβουμε ε, δράση για αυτό το θέμα αυτό στη εκθέσει για τον ανταγωνισμό. Τώρα για την Google, η ταχύτητα κάποιων ερευνών. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σε δέκα δευτερόλεπτα πρέπει να τελειώσετε, λέει ο πρόεδρος. Πιστεύετε ότι πρέπει να ε, ε, εξισορροπήσουμε την ταχύτητα της έρευνας με την ανάγκη ε, να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των επιχειρήσεων. Για την Google είπατε ότι ε, ε, θα έρθουν και άλλες υποθέσεις antitrust. Ίσως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε ποιες είναι αυτές. Και για το shopping ακούω ότι κάποιοι δεν είναι ικανοποιημένοι από το μηχανισμό που προσφέρετε. Εσείς καλύπτεστε από αυτό. Καταρχήν, για να απαντήσω στην Κέιτ και την ερώτηση για την ΕΚΤ, είπα ότι θα επανέλθω, ένα πράγμα που πρέπει να έχετε υπόψη είναι ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να ε, επενδύσουν με βάση τα δεδομένα της αγοράς, με τους όρους της αγοράς. Αυτό μπορεί να γίνει. Ποιοι είναι όμως οι όροι της αγοράς. Είχαμε αρκετέ περιπτώσει όπου έρχονται οι κυβερνήσει και λένε ότι θέλουμε να κάνουμε επενδύσει με όρου αγορά. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε σχετική απόφαση για να μην έχουμε πρόβλημα με κρατικέ ενισχύσει αργότερα. Και καμιά φορά αυτέ οι υποθέσει περιπλέκονται πολύ. Γιατί οι όροι τη αγορά δεν είναι αναγκαστικά 2 ή 3%. Εάν υπάρχει κίνδυνος, τότε τα επιτόκια θα είναι πολύ ψηλότερα. Και αυτό μπορεί να συμβεί επίσης. Οπότε υπάρχουν διαφορετικά διακυβεύματα εδώ όταν βλέπουμε κυβερνήσεις να αγοράζουν ομόλογα ε, από κάπου. Εξαρτάται από το πώς θα γίνει αυτό. Από την πλευρά της ΕΚΤ, όπως είπα, δεν μπορώ να απαντήσω. Τώρα, το... τα μέτρα αντιτράστ. Υπάρχει μια συμμετρία, διότι όταν κάνουμε έλεγχο συγχωνεύσεων, έχουμε ευθυγράμμιση συμφερόντων όταν πρόκειται για τον καθαρισμό του χρονικού ορίζοντα. Βέβαια, η εταιρεία μπορεί να θέλει να προχωρήσει συγχώνευση. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε ότι δεν θα ε, ζημιωθεί ο ανταγωνισμός. Το κοινό είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα και οι εταιρείες θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, ούτως ώστε να προχωρήσει η συγχώνευση το ταχύτερο δυνατό. Η ασύμμετρία συμβαίνει όταν γίνεται ας για ένα καρτέλ. Εκεί τα μέρη δεν θέλουν τόσο πολύ να συνεργάζονται, διότι εμείς κάνουμε έρευνα σε ένα μυστικό καρτέλ και μπορεί να υπάρξει πρόστιμο. Ε, είχαμε περίπτωση ε, προστίμου ύψους 4 δις ευρώ. Οπότε η απροθυμία τους να συνεργαστούν να ε, δώσουν αυτά που χρειαζόμαστε, ε, να απαντήσουν το ταχύτερο δυνατόν στο αίτημα για πληροφορία δεν είναι ίδιο όπως στην περίπτωση μιας διαδικασίας συγχώνευσης. Και εκεί είναι η δυσκολία το να δουλέψουμε με προθεσμίες. Και είναι πολύ σημαντικό, επειδή είμαστε ένωση κρατών δικαίου, είναι δύσκολο να ε, φροντίσουμε πάντα ε, ώστε να μπορούν να προσφύζουν τα συμφέροντά τους οι εταιρείε. Σίγουρα πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Η πρόσβαση στους φακέλους θα πρέπει να διευκολύνεται, πρέπει να είναι εύκολη. Διότι όταν στέλνουμε ας πούμε δήλωση ε, ένστασης, θα πρέπει η εταιρεία να βλέπει τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουμε εμείς εναντίον τους και αυτό θα πρέπει να γίνεται με αποτελεσματικό και σωστό τρόπο. Όλη η διαδικασία θα διευκολύνεται έτσι γενικότερα. Σίγουρα αυτό είναι μια πρόκληση και ένα πρόβλημα για τον προϋπολογισμό μας, γιατί θέλουμε πληροφοριακά συστήματα, πρέπει να έχουμε ανθρώπους ε, ε, ειδικού που ε, δεν τους είχαμε πριν από 5-10 χρόνια και να επενδύσουμε στα εργαλεία που διαθέτουμε για να επιταχύνουμε τις ερευνητικές διαδικασίες. Ε, στην περίπτωση Google είχαμε 5,2 terabytes δεδομένων για να τα δούμε. Παίρνει πολύ χρόνο. Πρέπει να έχουμε δηλαδή και τα απαραίτητα εργαλεία για την επεξεργασία τόσων πολλών δεδομένων. Αυτό είναι υψηλή προτεραιότητα. Δεν νομίζω ότι η απάντηση στο πρόβλημα είναι η προθεσμίας. Θα πρέπει οι πόροι να επενδύονται σωστά σε καλές διαδικασίες και εργαλεία. Τέλος, ε, ε, ε, έχω συναντήσει πολλούς που είχαν πρόβλημα με την Google και του συνάντησα για να ακούσω τη δική τους άποψη. Εμείς έχουμε επαφή με την αγορά. Ακόμα δεν έχουμε λάβει απόφαση για το θέμα της Google, αλλά παρακολουθούμε από κοντά. Γιατί δεν είναι το θέμα του, ε, της δημοπρασίας ε, καθ' αυτής, αλλά το πώς λειτουργεί αυτή. Και γι' αυτό αξιοποιούμε τους ε, τεχνικούς ειδικούς, εξετάζουμε και οι ίδιοι και είμαστε σε επαφή και με τους παίκτες στην αγορά. κυρία Λόπες Περμέχο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέει η κυρία Λόπερ Μπερμέχο για την παρουσία σας εδώ και την ε, διαθεσιμότητά σας. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα ήθελα να θέσω γύρω από τη γεωργία και από την ενέργεια. Στην περίπτωση της γεωργίας τα τελευταία χρόνια, χάρη ακριβώς και στην πίεση του Κοινοβουλίου, έχουν δημιουργηθεί κάποια, θα έλεγα, κάποιες μέθοδοι παρακολούθησης των τιμών που επιτρέπουν να γίνεται ε, μια σωστή ανάλυση της λειτουργίας της αγοράς τροφίμων. Και φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες μορφές καταχρήσης στον τομέα της ε, αγοράς αυτής, ιδιαίτερα από πλευράς των μεγάλων επιχειρήσεων που αγοράζουν το γεωργικό προϊόν και τελικά οι οργανώσεις των παραγωγών ε, βρίσκονται χωρίς άμυνες και πληρώνουν το τίμημα. Διαρωτώ με λοιπόν εσείς σκέφτεστε να αλλάξετε τις ισχύουσες οδηγίες έτσι ώστε και η πολιτική του ανταγωνισμού στον τομέα της γεωργίας να εφαρμοστεί με πράγματι ενιαίο και δίκαιο τρόπο και μπορεί να υπάρξουν ρυθμίσεις στα πλαίσια της ΚΑΠ για να προστατευθούν τα συμφέροντα των γεωργών. Τώρα, για να αναφερθούμε στο θέμα αυτό, αναφερόμαστε βέβαια και στην συγχώνευση Μπάγερ Μονσάντο. Τώρα σε έναν άλλο τομέα φαίνεται ότι η βοήθεια στις ανανεώσιμες πήγες ε, γενικά δεν επιδοτούνται πλέον και έχουν υπάρξει και αποζημιώσεις από τις ε, διάφορες χώρες προς τις εταιρείες που είχαν επενδύσει στο παρελθόν στον τομέα αυτό. είναι κάτι το οποίο ευνοεί φυσικά τις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι κάτι το οποίο δεν βοηθά τις ανανεώσιμες πηγές και φαίνεται ότι γενικά οι αντιστάσεις της αγοράς καυσίμων είναι αυτό το οποίο μας εμποδίζει κυρίως για να περάσουμε σε μια πραγματική νέα ανοιχτή αγορά με ανανεώσιμες πηγές. Όλοι αυτοί οι τομείς έχουν πολύ μεγάλη σημασία γιατί αφορούν την καθημερινότητά μας. Το πρωί ξυπνάς, φτιάχνεις ένα καφέ, οπότε χρειάζεσαι την ενέργεια και τη γεωργία για να το κάνεις αυτό. Uh, Έχουμε ξεκινήσει κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα μας δώσουν την δυνατότητα να ενισχύσουμε το κομμάτι της παραγωγής. Θα πρέπει να γίνει πιο λειτουργική η προσπάθεια αυτή. Σαν παράδειγμα για τις αρρώσιμες γεές σε διάφορα προϊόντα όπως τα έλαια και τα λοιπά θα πρέπει να διευκολύνουμε τους παραγωγούς να συνεργαστούν να δημιουργήσουν όχι μόνο μονοπόλια αλλά αποτελεσματικές ομάδες προώθησης και πώλησης των προϊόντων τους. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε να δουλέψουν αυτές οι προσπάθειες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες τέτοιες προσπάθειες είναι πραγματικά ευεργετικές για τους παραγωγούς. Τώρα για τα θέματα των εγγυημένων εισοδημάτων είναι κάτι το οποίο συζητάμε στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων για την ΚΑΠ. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το συζητήσει στο μέλλον το θέμα αυτό. Ο συνάδελφος Χόγκαν φυσικά είναι ο αρμόδιος επίτροπος για να το συζητήσει. Πάντως στην παρούσα φάση βρισκόμαστε και στην εξέταση της διαδικασίας συγχώνευσης Bayer και Μονσάντο. Θα πρέπει ε, να, να μην παραγνωρίσουμε το ότι ανεξάρτητα από την ε, συγχώνευση οι γεωργοί χρειάζονται επιλογή, να επιλέξουν τη σπορία, να επιλέξουν τα ζυζανιοκτώνα, να έχουν δυνατότητες επιλογής και να βελτιώνεται η κατάσταση γιατί χρειαζόμαστε σαν παράδειγμα ζυζανιοκτώνα τα οποία να μην είναι τόσο βλαπτικά για το περιβάλλον, ε, χρειαζόμαστε ε, σπόρους οι οποίοι να είναι αποδοτικότεροι και οικονομικότεροι και να επιτρέπουν στους γεωργούς να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα στον τομέα αυτό ε, τώρα των συγχωνεύσεων ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί οι κανόνες υπάρχουν, οι γενικοί κανόνες υπάρχουν έτσι ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον και να προστατευθούν οι ε, καταναλωτές από τα ζυζανιοκτώνα και γενικότερα από τις αρνητικές πιθανώς επιπτώσεις. Διερευνούμε επίσης ορισμένες περιπτώσεις όταν υπάρχουν ανησυχίες για τις τιμές, όταν πράγματι κάποιοι πολύ μεγάλοι αγοραστές μπορεί να στρεβλώνουν τις αγορές. Έχουμε την περίπτωση της μεγάλης ζηθοποιίας Interbrew. Επίσης πρέπει να βοηθήσουμε τους γεωργούς να φτάνουν τα προϊόντα τους στα ράφια των επιχειρήσεων Ε, μερικές φορές είχαμε περιπτώσεις στη Γαλλία σαν παράδειγμα προώθησης των γαλλικών προϊόντων ε, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα σε ορισμένους τομείς. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε λοιπόν τέτοιες καταστάσεις και δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πόλεμο για το ποια είναι τα προϊόντα που θα φτάσουν στα ράφια γιατί κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο λαμβάνονται οι μη αντίμετρα. Αν τα προϊόντα μου δεν φτάνουν στα δικά σου ράφια ούτε και τα δικά σου θα φτάνουν στα δικά μου στη συνέχεια και αυτό θα καταστήσει την κατάσταση των γεωργών ακόμα πιο δύσκολη και φυσικά οι επιλογές των πολιτών θα είναι πολύ μικρότερες. Στον τομέα της ενέργειας τώρα ε, κοιτάξτε, εδώ μπορούμε να συζητήσουμε για ώρες για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την αγορά ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε σε μία μεταβατική φάση και η μεταβατική αυτή φάση θα κρατήσει αρκετά χρόνια. Έχουμε μία βαριά κληρονομιά θα έλεγα και με τους παραδοσιακούς τομείς παραγωγής και με την πυρηνική ενέργεια και με τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα, στα κρατη κράτη-μέλη. Ε, σε πολλές ε, χώρες ε, υπάρχουν στον τομέα της ενέργειας και σοβαροί κίνδυνοι blackout. Υπάρχει μια ευαισθησία ως προς αυτό, οπότε υπάρχει και ανάγκη δημιουργίας ε, μηχανισμών προστασίας, αν θέλετε, τα backup mechanisms, οι αναπλήρωσης. Και θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί αυτοί οι οποίοι μπορεί να, ενσωματωθούν, να ενσωματωθούν στις αγορές. Θα πρέπει οι μηχανισμοί αυτοί να είναι ανοιχτοί φυσικά και σε επίπεδο διαμεθοριακής συνεργασίας. Θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά και θα πρέπει επίσης να επιτρέψουμε και στις ανανεώσιμες πηγές να συμμετέχουν στους μηχανισμούς αυτούς. Ιδιαίτερα το διαμεθοριακό κομμάτι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί αν θέλει κανείς μια ενεργειακή ένωση τότε η διαμεθοριακή συνεργασία είναι κομβική. Τώρα υπάρχουν ε, κάποιες διαφορές ανάμεσα στα μέτρα τα οποία ισχύουν, αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές επιλογές του energy mix που χρησιμοποιεί και αποφάσισε στο παρελθόν κάθε χώρα. Πάντως βασίζεται σε μια αποδεδειγμένη ανάγκη να υπάρχει ένας μηχανισμός προστασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και αυτό θα μας επιτρέψει σιγά σιγά να περάσουμε σε ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας το οποίο θα είναι συμβατό με τα, με τις περιβαλλοντικές μας ανησυχίες. Κυρία Σκορτκατώ, είμαι Βρετανίδα, προέρχομαι από νοτιοανατολική Αγγλία με πολλές θέσεις εργασίας. Ο κύριος Δραγκη μας είπε ότι εκτός της εσωτερικής αγοράς οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις της Βρετανίας δεν θα έχουν το δικαίωμα να ε, συναλλάσσονται ελεύθερα με ευρωπαϊκέ αντίστοιχε ε, των κρατών μελών, γιατί θα έχουν χάσει τα πιστοποιητικά του. Δεν με βέβαια, γιατί το, περί... το και ο κύριο Μπαρνί, το κατέστησε απόλυτο σαφέ, λέγοντα ότι δεν θα υπάρχει φιλόδοξη εταιρική σχέση χωρί κοινό πεδίο για τις κρατικές ενισχύσεις, ε, του ανταγωνισμού, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, τους κανόνες για, την, για τα τρόφιμα. Αυτό σημαίνει προ, προδιαγραφές υγείας, περιβάλλοντος, χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς μαζί του. Ε, προς τα τέλη του προηγούμενου μήνα κάνατε μια έρευνα για, την, ε, για τις φορολογικές αιρέσεις από εταιρείε που ανήκουν στο Βρετανικό κράτος έχει από ό,τι φαίνεται διαπιστωθεί παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, αθέμητος δηλαδή ανταγωνισμός φορολογικός από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συνέπεια αυτής της έρευνας νομίζω θα είναι ορατή λίγο πριν, να, ή αισθητή λίγο πριν να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αμέσως μετά. Επομένως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις δηλώσεις για μια βαθιά και ιδιαίτερη σχέση που θέλει και η Πρωθυπουργό εννοεί ότι πρέπει να τηρεί τους ίδιους φορολογικούς κανόνες του Ηνωμένου Βασίλειο με τα υπόλοιπα 27 κράτη που μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι υπεράκτιες επίσης ε, κτίσεις της, του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπουν σε κατάλογο παραδείσων φορολογικών, ε, σε μαύρη λίστα. Ε, θα επιβάλλεται, θα με αυστηρούς κανόνες η συμμόρφωση στο ευρωπαϊκό δίκαιο, το φορολογικό και λοιπό και κυρίως σε σχέση με τις παράκτιες ε, κτίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Απάντηση. Όπως είπατε, δεν διαφωνεί κανείς με τον Παρνιέ. Ναι, και είναι λογική είναι έτσι. Ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού ίσον ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Και για τις ίδιες τις βρετανικές επιχειρήσεις καλό είναι να μην βρίσκονται σε σχέση του ανταγωνισμού όταν είναι σε σχέση ανταγωνισμού με επιχειρήσεις της υπόλοιπης Ευρώπης. Άρα λοιπόν μια απλή και ρεαλιστική θέση προς το συμφέρον όλων ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και γι' αυτό και με πολύ μεγάλη σαφήνεια εξετέθη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Απρίλιο ότι αυτή είναι η εντολή για τη διαπραγμάτευση τη συμφωνία για το Brexit. Ξεκινήσαμε την έρευνα για την εξαίρεση του ομίλου του χρηματοπιστωτικού, γιατί υπάρχουν λόγια ανησυχία. Και για πολύ σοβαρούς λόγους έχει προβλεφθεί η εξαίρεση στη σχετική νομοθεσία. Αυτό καταρχάς μας έβαλε στις σκέψεις και όταν κάναμε τις προκατακτικές έρευνες άρχισαμε να ανησυχούμε κιόλα. Χρειάστηκε βέβαια σε πολύ στο διάστημα να βρούμε τα στοιχεία μέχρι να ολοκληρωθεί το Brexit. Πρέπει να είμαστε και εμείς έτοιμοι. Θα δούμε βεβαίως αν θα τα καταφέρουμε. και δεν γνωρίζω ποιο θα μπει στον κατάλογο των φορολογικών ε, παραδείσων. Ο συνάδελφο Μοσκοβισή είναι αρμόδιο. Και ξέρετε ότι κάνουν εντατική δουλειά για να προλάβουν ε, τη δημοσίευση πριν από τα Χριστούγεννα συγκεκριμένες γνώσεις για το πώς προχωρεί αυτή η υπόθεση δεν έχω και ω εκ δεν μπορώ να απαντήσω στη δεύτερη ερώτησή σα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άνιμανς. Θα μιλήσω στα Ολλανδικά, αν μου επιτρέπετε. Μια ερώτηση για τα Paradise Papers. Στις 11 Νοεμβρίου δώσατε μια συνέντευξη, παραθέτω τι είπατε. Πρέπει να πω ότι αυτό ήταν ηλεκτρικό σοκ και έτσι θα επιταχυνθούν οι αποφάσεις από το Συμβούλιο τέλος του παραθέματος. Τώρα έχουν γίνει πολλές αποκαλύψεις για τα Paradise Papers και φαίνεται ότι οι φορολογικές αρχές του Βελγίου είχαν επαφές με βρετανικές εταιρείες offshore. Αυτά τα γνωρίζετε. Τα έχετε υπόψη. Και ε, αφαιρθήκατε και εκεί όταν είπατε ότι ήταν ένα ηλεκτροσόκ, τα Paradise Papers και θα ξεκινήσετε διαδικασίες κατά του Βελγίου, όπως και κατά των πολυεθνικών, γιατί και οι Βέλγοι πολίτες ε, ε, άκουσα με μεγάλη δυσφορία όλα αυτά. για όλες αυτές τις ε, δραστηριότητες. Είναι πολύ νωρίς να πούμε αν θα με διαδικασίες συγκεκριμένες. Τώρα επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες από τα Paradise Papers και αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας, τότε θα ξεκινήσουμε νέες διαδικασίες. Ε, χρησιμοποίησα έντονη γλώσσα, γιατί θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει οι πολίτες να ε, βλέπουν ότι όλες οι εταιρείε και όχι πολλές πληρώνουν φόρους. Πολλοί είναι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες είναι σε μια εθνική ε, ε, επιχείρηση, σε μια ε, εταιρεία. Βλέπουν ότι δίνει μάχη καμιά φορά για να παραμείνει στην αγορά. Καμιά φορά ανταγωνίζεται εθνικές που είναι οργανωμένες πολλές φορές με τρόπο που τους επιτρέπει να ελαχιστοποιούν τους φόρους που πληρώνουν. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι θέμα ίσων κανόνων ανταγωνισμού, είναι και θέμα κοινωνικού συμβολέου, αν θέλετε, για το πώς ε, δραστηριοποιείται κάποιος επιχειρηματικά σε μια κοινωνία όπου χρειάζεται ε, δρόμους, πελάτες ε, και η κοινωνία θα πρέπει να μπορεί να επενδύει στην υγεία, την παιδεία, στις υποδομές για να υπάρχει δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει για να δούμε, ορίστε, δεν ξέρω, ε, δεν ξέρω αν ε, πέρασε το μήνυμα ή ε, Βρετανική κυβέρνηση συμμετέχει σε προγράμματα συνεργασίας με τα τις Παρθένους νήσους. Το Βέλγι, οι Βέλγοι πολίτες έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ και βεβαίως στο Συμβούλιο μπορείτε να ανακαλέσετε στην τάξη το Βέλγιο. Εντάξει, τότε θα ξαναπώ αυτό που είπα στην αρχή. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε. Εμείς ε, εξετάζουμε διεξοδικά τα στοιχεία. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Διότι όλοι έχουν το δικαίωμα της αμφιβολίας, στο τεκμήριο αθεότητας και ε, η συζήτηση έγινε στο Βελγικό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι κάνατε την ερώτηση και πήρατε και την απάντησή σας. Ο κύριος Χέις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ε, καλωσορίζω για μια ακόμη φορά Επίτροπε. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα την εκλογική μου περιφέρεια είναι το θέμα των Ιρλανδικών τραπεζών που ασχολήθηκαν με τα σκάνδαλα με τις υποθήκες στο παρελθόν. Πάρα πολλοί Ιρλανδοί πολίτες και κάτοχοι υποθήκων έχασαν γενικά τα περιουσιακά του στοιχεία, αναγκάστηκαν να πληρώσουν επιπλέον χρήματα. Τα θέματα αυτά εξετάστηκαν από την Ιρλανδική Κεντρική Τράπεζα και θα ήθελα να μάθω αν υπήρξε δραστηριότητα τύπου καρτέλ από τα Ιρλανδικά πιστοτικά ιδρύματα. Υπήρξε μια στρέβλωση της τραπεζικής αγοράς στην Ιρλανδία. Στις 25 Οκτωβρίου έστειλα μια επιστολή στη Γενική σας Διεύθυνση και αναφέρθηκα σε δύο παραδείγματα Αυστραλιανών τραπεζών και άλλα παραδείγματα στα οποία η γενική σας διεύθυνση είχε ασχοληθεί με θέματα παραγόγων και πήρα μια απάντηση από πλευρά σας αυτή την εβδομάδα σχετικά με τους ισχυρισμούς τους οποίους είχα διατυπώσει. Λέτε ότι εξακολουθείτε να εξετάζετε την κατάσταση την οποία έχω περιγράψει Λέτε επίσης ότι το θέμα αυτό είναι Ιρλανδικό και ότι θα ήταν καλό ε, να ασχοληθεί με το θέμα αυτό η Ιρλανδική Αρχή επί του ανταγωνισμού. Ε, αναρωτιέμαι, για αυτές τις τράπεζες ε, είναι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υπεύθυνο το SSM γύρω από τις τράπεζες αυτές. Οπότε λοιπόν διαρωτώ με, τι ακριβώς επιθυμείτε, θέλετε επιπλέον αποδείξεις από αυτούς οι οποίοι υπέστησαν ζημίες, θέλετε να σας στείλουν επιπλέον στοιχεία στη γενική σας διεύθυνση. Είναι ένα τρομερό σκάνδαλο τοπικά και νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε την αλήθεια και στα πλαίσια του τομέα του ανταγωνισμού και εδώ έχετε τις δυνατότητες να το κάνετε εσείς ειδικά. Όπως είπατε, αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Είναι θέματα τα οποία επηρεάζουν μεμονωμένες πολίτες, ε, οικογένειες, τις υποθήκες τους, τα δάνειά τους, τα στεγαστικά, τα οποία τους κοστίζουν πάρα πολλές φορές ε, πάρα πολύ και είναι σημαντικό βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ε, τα ένα από τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Ένα από τα σημαντικά θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε επίσης είναι κάθε φορά η έρευνα να γίνεται από την αρχή η οποία είναι στην καλύτερη αν θέλετε θέση. Το θέμα δεν είναι ότι δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε κάτι, αντίθετα. Το θέμα είναι να βρούμε το ποιος μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο πράγμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον πιο γρήγορο τρόπο και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και αυτό το οποίο εμείς, εμείς αναζητούμε είναι οι επιπτώσεις στις αγορές. Ανεξάρτητα αν είναι Ευρωπαίοι εταίροι ή παγκόσμιοι εταίροι, μας ενδιαφέρει το πώς λειτουργούν οι αγορές. Στο εσωτερικό της Ευρώπης υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αγορές. Υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις, υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες διαμόρφωσης της αγοράς υποθηκών ή της αγοράς στεγαστικών δανείων, αν θέλετε. Συνεπώς λοιπόν είναι σαφές ότι θα πρέπει να εργαστεί για το θέμα αυτό η αρμόδια Ιρλανδική Αρχή επί του ανταγωνισμού η οποία έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες τις οποίες όλοι χρειαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια αν κάποιος λέει σε μια φάση ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά ε, και θα ήθελα να προειδοποιήσω για τις εξελίξεις αυτές δεν ξέρω αν χρειάζεται να προηγηθεί κάτι τέτοιο έτσι ώστε να κινητοποιηθεί αν θέλετε μετά από συγκεκριμένη καταγγελία η αρμόδια επί του, ε, επί του ανταγωνισμού αρχή. Πάντως υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήσει κανείς με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής ακόμα και ανώνυμα ε, υπάρχουν στοιχεία λοιπόν τα οποία απαιτείται και τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μια έρευνα είτε από δικής μας πλευράς είτε από πλευράς των εθνικών αρχών. Θα συνεχίσουμε εμείς να ελέγχουμε τις αγορές αυτές μετά από τη χρηματοπιστωτική κρίση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η αγορά η τραπεζική. Έχουν υπάρξει νομοθετικές ρυθμίσεις για να καταστήσουμε πιο ασφαλή, πιο προβλέψιμη και ίσως και λίγο πιο βαρετή την χρηματοπιστωτική αγορά γενικότερα, αλλά αυτό είναι ο στόχος μας και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε από κοντά τις εξελίξεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ζητούσα από οιονδήποτε, ο οποίος θεωρεί ότι έχει αποδείξει σε σχέση με τον τομέα του ανταγωνισμού γύρω από αυτήν την υπόθεση, να μας ενημερώσει με τον, ένα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φυσικά εμείς μπορούμε να λειτουργήσουμε απόρριτα, μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας και εκεί θα δούμε πού είναι το καλύτερο επίπεδο αναζήτησης στοιχείων και επίλυσης τελικά του προβλήματος. Ευχαριστώ, Μπορτζάνη. Συμπορτζάνη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, επιτρέψτε μου να συνεχίσω στην ίδια κατεύθυνση γεωργικά θέματα είχαμε πριν από λίγο, σε αυτά θα μείνω. Ίσως να είστε ενήμεροι ότι στην Επιτροπή Γεωργίας και γενικά στις εξωτερικές της δράσεις υπάρχει συναντήληψη πως οι συλλογικέ δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους ε, και ο προγραμματισμός ε, της παραγωγής και τα συμβόλαια πωλήσεων είναι απαραίτητα τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία της κοινή γεωργικής πολιτικής, τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα θα έπρεπε να αποκλείονται από την εφαρμογή του περιφήμου άρθρου 101 της συνθήκης. Βεβαίω, ε, πρέπει να γίνονται ε, γνήσια κοινέ δραστηριότητε που συμβάλλουν στην ε, παροχή τη υπηρεσία των γεωργών. Επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρχε δυνατότητα για παρεκκλήσεις που δεν είχε αξιοποιηθεί πλήρως, γιατί δεν ήταν απολύτως σαφείς αυτές οι παρεκκλήσεις και υπήρχαν δυσκολίες ω προς την εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού που δεν έδωσαν τις παρεκκλήσεις στους γεωργούς, γιατί δεν ήταν βέβαιες αν μπορούσαν να το πράξουν. Χαιρόμαστε λοιπόν που ο κανονισμό όπνης τους μπορεί να απλοποιήσει τους κανόνες για τις ενώσεις και οργανώσεις των παραγωγών, το ρόλο και τις αρμοδιότητες αυτών. Επιπλέον, επικρατεί η πεποίθηση ότι ο ιδιάζων χαρακτήρας της, ε, του γεωργικού τομέα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και στην πολιτική του ανταγωνισμού. Αυτό ήταν και το νόημα του μηνύματος κυρίου Σάντ εξάλλου. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας και θα ήθελα τα σχόλιά σας. Κύριε Φεστάκερ ε, όντως είναι δύσκολο να τοποθετηθώ σε σχέση με τις προτινόμενες ε, αλλαγές, διότι δεν έχει γίνει αξιολόγηση επιπτώσεων. Άρα δεν μπορώ να γνωρίζω πώς θα λειτουργήσει το σύστημα, αν θα πλουστεύσει τα πράγματα. Γιατί έχουμε κάνει προσπάθεια υπό τον πρόεδρο Γιουνκέρ, αλλά και υπό τον πρώτο πρόεδρο Φραντ Τίμερμανς, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή νομοθεσία, το καλύτερο δυνατό νομοθετικό έργο και να ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα φέρει το κάθε νομοθέτημα. Γιατί αυτό ε, το πράττουμε και για λόγους σεβασμού προς τον νομοθέτη. Στις αλλαγές λοιπόν, τις σχετικές ε, με τον κανονισμό Omnibus, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, διότι δεν έχει γίνει αξιολόγηση επιπτώσεων, δεν έχει γίνει δημόσια διαβούλευση. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι και να δηλώσουμε ότι μπορεί να αποβεί ισόφελος των μικρότερων παραγωγών, όφελο του κάθε καταναλωτή, γιατί δεν είμαστε βέβαιοι ότι αυτός είναι ο τρόπος να εξασφαλιστεί για τον Γεωργό ε, μεγαλύτερη δυνατότητα δράσης στην αλυσίδα παραγωγής προσθεμένης αξίας. Αυτό το είπα και νωρίτερα στην κυρία Λόπες ότι είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη θέση του παραγωγού να του δώσουμε μεγαλύτερη αξία και εξουσίες στην αλυσίδα παραγωγής προσθέμενης αξίας, χωρίς όμως να είναι και να μένουν με δεμένα τα χέρια, να μπορούν να έχουν αναλλακτικέ. Θα πρέπει οι ίδιοι να μπορούν να αποφασίσουν τι θα θέλουν να κάνουν και πώς. Και είναι πολύ περιορισμένος ο ρόλος στην νομοθεσία για τις αρχές ανταγωνισμού που θα μπορούσαν να προστατεύουν αυτή την ευχέρεια επιλογών. Είχαμε στο παρελθόν περιπτώσεις όπου ήταν πολύ δύσκολο παραγωγός που είχε μια διαφορετική ιδέα, μια διαφορετική φιλοδοξία. Ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό ή με διαφορετικό τρόπο, να ε, ιδρύσει μια δική του φερρυπίν οργάνωση ή ένωση παραγωγών, γιατί δίπλα υπήρχε ένας τιτάνας, μια μεγάλη οργάνωση παραγωγών και δεν είχε περιθώριο δράσης. Και εκεί θα έπρεπε να μπορούν οι αρχές συνταγωνισμού να παρεμβαίνουν και βεβαίω όταν λαμβάνονται αποφάσει από τον νομοθέτη τι σέβομαι, αλλά δυστυχώ δεν είμαι σε θέση να δώσω απάντηση στην ερώτηση αν αυτό αποτελεί απλοποίηση, αν μπορεί να φέρει αποτελέσματα, αν μπορεί να φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και για την προστασία του παραγωγού αλλά και για την εξασφάλιση της δυνατότητα για αυτόν να δημιουργήσει μια νέα οργάνωση ένωση εάν θεωρεί ότι δεν τον ικανοποιεί αυτή στην οποία ανήκει. Και αυτό το λέω ανησυχία και πάντως με κάθε σεβασμό στις ε, επιλογές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον τριμερή διάλογο. Αλλά ενώ εμείς αποτελούμαστε σε μια προσπάθεια ώστε να υπάρχει δημόσια διαβούλευση, αξιολόγηση των επιπτώσεων μιας προτινόμενης ε, προ, ιδέας ε, πράξης ομοθετικής που θα σας καταθέσουμε για να είμαστε βέβαιοι ότι θα ε, φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους πολίτες που θέλουμε να ενισχύσουμε. Ευχαριστώ Μαρτουσέλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από δέκα περίπου μήνες ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια έκθεση με 183 συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω την Επιτροπή. Πόσες από αυτές τις συστάσεις λάβατε υπόψη και ποιες. Διότι σήμερα η Επιτροπή ετοιμάζεται να συζητήσει μια νέα ετήσια έκθεση για τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να αντιληφθώ, εάν απλώ χάνουμε το χρόνο μα, γιατί δεν, σας, ε, δεν τις λαμβάνετε υπόψη αυτέ τι ε, εκθέσει και τι συστάσει, ή όχι. Μπορείτε να μας πείτε 183 σημεία και συστάσει. πόσα και ποια από αυτά ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή. Δεύτερη ερώτηση. Στην Ιταλία γίνεται συζήτηση για την αρμοδιότητα για ανάληψη νομοθετικού έργου σε σχέση με τα θέρετρα. Έχει κάνει μία πρόταση κυβέρνηση νομοθετική, ορισμένες ε, όμως περιφέρειες στην Ιταλία να λαμβάνουν πρωτοβουλία μονομερός γιατί θεωρούν ότι είναι περιφερειακή αρμοδιότητα. Μπορείτε εσείς από τη δική σας θέση να μας πείτε ποιος θα είχε αρμοδιότητα, κράτος ή περιφέρεια. Γιατί κινδυνεύουμε να περιέλθουμε σε μεγάλη νομοθετική ε, ασάφεια και σύγχυση. Θέλετε να μου πείτε ποιος τομέας ήταν ε, για τις ε, παρεκκλήσεις ε, που θα επέτρεπαν στις περιφέρειες να ρυθμίσουν το θέμα. Πρόκειται για τις παραχωρήσεις για εκμετάλλευση ακτών. Προχώρησε σε μια νομοθετική πράξη η κυβέρνηση, πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Κυρία Φερστάγκερ. Για την πρώτη ερώτηση, τον αριθμό των συστάσεων και αν τις ακολουθούμε ή αν εμπνεόμαστε από αυτές. Δεν είναι έτσι η δουλειά σε σχέση με τις ε, εκθέσεις για τον ανταγωνισμό, ε, γιατί αυτές οι εκθέσεις είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο ως τελικό προϊόν, αλλά και ως διαδικασία παραγωγής της έκθεσης. Γιατί έχουμε νομίζω πολύ στενή επαφή κατά τη διάρκεια της κατάρτισης έκθεσης με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές, έτσι ώστε και να γνωρίσουμε καλύτερα, τις, ε, να εξοικειωθούμε με τις ιδέες τους, τις ανησυχίες τους, τις προτεραιότητες, ε, τη διάθεσή τους. Και γι' αυτό δεν έχουμε ένα κατάλογο επιδόσεων που να λέμε ε, να η μία να η άλλη τις εφαρμόσαμε, γιατί έχουν και πολύ διαφορετική φύση αυτές οι συστάσεις. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν το ίδιο ειδικό βάρος. Ούτε θα ήθελα να πέσουμε στον πειρασμό να πούμε α, τις εύκολες τις θέτουμε σε εφαρμογή και τις άλλες τις αφήνουμε στην άκρη. Δεν είναι αυτός τρόπος συνεργασίας. η συνθήκη προβλέπει ένα συγκεκριμένο τρόπο συνεργασίας μεν, αλλά πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει σε μια μορφή συνεργασίας ουσιαστική που μας επιτρέπει πιο στενές σχέσεις ε, και με το Κοινοβούλιο, τα μέλη της δικής της Επιτροπής ε, και τους αρμόδιους για τον ανταγωνισμό που ουσιαστικά προβλέπει η συνθήκη και αυτό είναι πολύ θετικό γιατί μας επιτρέπει πιο στενή συνεργασία μαζί σας με εσάς που εκπροσωπείτε τους πολίτες. Βεβαίω, εάν σα ενδιαφέρει ιδιαίτερα, πολύ ευχαρίστω να σας στείλω μια γραπτή απάντηση. Αλλά θέλω να επισημάνω, να επιμείνω σε αυτό, ότι σε όλη τη διαδικασία παρακολουθούμε, ενστερνιζόμαστε, αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται από μας, τι μας ζητάτε. Και οπωσδήποτε ποτέ δεν είναι χαμένος σκόπος η προσπάθεια αυτή να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την επιβολή, την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού για το καλό των πολιτών στα κρατη Το πώς οργανώνουν το, στο εσωτερικό τους τις διαδικασίες στα κράτη-μέλη πάλι είναι δικό τους θέμα. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου είναι αποκεντρωμένη και η ε, συλλογή ε, των φόρων. Μπορεί να έχουν διαφορετικό δημοκρατικό τρόπο οργάνωσης ε, τα κράτη, πάντα βέβαια με το σεβασμό των θεμελιωδών αρχών του ανταγωνισμού. Αλλά προφανώς δεν χρειάζεται οι Βρυξέλλες να επιβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουν τα κράτη-μέλη ε, τη δομή του εσωτερικά, ούτε ως προς τις κρατικές επιδοτήσεις, ούτε ως προς τα άλλα ε, θέματα και τις δράσεις που έχουμε για να προστατεύουμε τους καταναλωτές και την αγορά. Ναι, αυτό ήταν σχετικό με την οδηγία Bolkenstein και την εφαρμογή της, το ερώτημα. Κυρία Γκίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε. Δύο θέματα, τα άλλα τα καλύψατε. Για τη φορολογία. Είπατε ότι οι κανόνες κρατικής ενίσχυσης ε, θα πρέπει να εξετάζονται σε βάση εξατομικευμένη και αυτό είναι πρόβλημα γιατί έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε δικαιότερο φορολογικό καθεστώς αν ρυθμίζουμε κατά περίσταση τα θέματα. Ένα παράδειγμα. Μιλήσατε και για τους φορολογικούς παραδείσους, blacklist κλπ. Καλό θα ήταν να έχουμε πιο διαρθρωμένη προσέγγιση στον τομέα των ε, ελέγχων. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και απαιτήσει ε, από τους πολίτες να δούμε το θέμα μέσα από το πρίσμα του ανταγωνισμού και να ε, διευκολύνουμε την κατάργηση φορολογικών παραδείσων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και πιο αυτόνομα τα φορολογικά καθεστώτα. Επίσης, οι μεγάλες εταιρείες πληροφορίας και ε, ε, και ο ρόλος που παίζουν στην παγκοσμιοποίηση. Βέβαια, είπατε ότι πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις για να λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Στις ΗΠΑ τώρα οι δημοκρατικοί ασχολούνται με αυτό το θέμα πολύ το κάνουν βασικό θέμα στην προεκλογική τους εκστρατεία, ότι πρέπει δηλαδή να υπάρχουν εργαλεία ανταγωνισμού που θα ελέγχουν τις ψηφιακέ εταιρείε. Αλλά και ε, στην Ανατολή βλέπουμε μεγάλες εταιρείε δεδομένων ε, ε, που έχουν ε, γίνει πολύ μεγαλύτερες εταιρείε ε, και στο Facebook θα πρέπει, βλέπετε ότι αυτοί προχώρησαν ένα βήμα περισσότερο από τους νομοθέτες που δεν πρόλαβαν να προσαρμοστούν. Αυτές οι ανάγκες θα, δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη και τι διαχωρισμοί πρέπει να γίνουν εκεί. Για το τελευταίο ερώτημα, νομίζω ότι η συμπεριφορά παίζει ρόλο, διότι είναι πολύ μεγάλη εταιρεία πρέπει να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Εάν σέβεται ουσιαστικά τον ανταγωνισμό, μπορούμε να έχουμε μία επιλογή. Εισόδου στην αγορά επένδυση σε καινοτομίε, παρουσίαση των καινοτομιών στους πελάτες. Πριν από 10 χρόνια αυτές οι εταιρείες δεν ήταν οι μεγαλύτερες εταιρείες ε, παγκοσμίω. Δεν ξέρουμε και πώ θα είναι η κατάσταση σε 10 χρόνια από τώρα. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό ε, είναι αυτό που συζητούσαμε και με τον κύριο Φέρμπερ πριν. Το πώς μια οικονομία που στηρίζεται σε δεδομένα επιτρέπει τον ανταγωνισμό. Αυτά όλα πρέπει να τα βλέπουμε ε, πολύ προσεκτικά. Ε, θα πρέπει η ύπαρξη των πολλών δεδομένων να μην αποτελεί εμπόδιο στην είσοδο στην αγορά. Η συμπεριφορά στην αγορά είναι σημαντική για να φροντίσουμε ότι θα παραμείνει ανοιχτή η αγορά. Και είναι ένα παράδοξο ότι για να έχουμε ανοιχτές αγορές θα πρέπει να παρεμβαίνουμε. Διότι αν δεν παρέμβουμε στην αγορά, ο κίνδυνος είναι να κλείσει η αγορά και στο τέλος να έχουμε μόνο μονοπόλια. Και αυτά θα εξυπηρετούν όπως νομίζουν καλύτερα εκείνα την αγορά. Τώρα, ένα δίκαιο φορολογικό καθεστώς. Ναι, δεν γίνεται αυτό με κατά περίπτωση εξέταση των κρατικών ενισχύσεων. Αυτό είναι μέρος της λύσης. Γι' αυτό η Κομισιόν έκανε αυτή τη συνολική προσέγγιση για να αντιμετωπίσει το θέμα με τρόπο διαρθρωμένο, όπως είπατε και εσείς. Γιατί σε περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων ε, σίγουρα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξουν επιλεκτικές, ε, επιλεκτικά ωφέλη και πλεονεκτήματα, να τηρήσουμε τις συνθήκες. Ε, η περίπτωση της Fiat δεν μπορεί να επαναληφθεί γιατί το Λουξεμβούργο άλλαξε τους κανόνες χρηματοδότησης των εταιριών, στην Κύπρο έγινε το ίδιο, άλλαξαν οι κανόνες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, στην Ιρλανδία άλλαξαν τους κανόνες για τις ε, διπλές Ιρλανδικές δομές, οπότε αλλάζουν τα κράτη-μέλη με δική τους πρωτοβουλία τους κανόνες τους και έχουμε αυτή, αυτή τη διαρθρωμένη προσέγγιση και αυτό αντικατοπτρίζεται στην νομοθεσία που προτείνει ο κ. Μοσκοβισή. Ε, βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να τα διευκολύνουμε γιατί αυτά τα προγράμματα είναι πάρα πολύ σύνθετα. Δεν ε, καταρτίζονται μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ε, ε, επηρεάζονται από τους ειδικού σε φορολογικά θέματα κλπ. Και εμείς θα πρέπει να αφυπνίσουμε τις ε, αρμόδιες αρχές για να ασχοληθούν με μια επιθετική φοροαποφυγή, για παράδειγμα. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια και ειλικρίνεια. Και εδώ όντως έχουμε μια διαρθρωμένη προσέγγιση. Σίγουρα κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί μας για να γίνουν όλα αυτά. Και έχουν γίνει πολλά περισσότερα τα τελευταία τρία χρόνια από αυτά που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Και ακόμα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Γιατί υπάρχουν ε, νομοθετικές προτάσεις που δεν έχουν ακόμη ε, εγκριθεί Ε, για τον, ε, την ενιαία φορολογική βάση για τις εταιρείες. Επίσης χρειάζονται ε, αναφορές αναχώρα για να βοηθήσουμε στη διαφάνεια και την αλλαγή. Και το καλό με τις διαρροές είναι ότι δείχνουν ότι αλλάζουν τα πράγματα. Θα έρθουν και άλλες διαρροές νομίζω. Οι πολίτες ε, θα αρχίσουν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει αλλά οι διαρροές θα καταδείξουν τις αλλαγές που χρειάζονται. Ένα θέμα που δεν έχει συζητηθεί όμως πολύ είναι η εφαρμογή. Γιατί η θέσπιση νομοθεσίας είναι ένα πράγμα, αλλά στην πράξη θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Οι φορολογικές αρχές σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν τους πόρους, τις ικανότητες τις προσλήψεις, να κάνουν τις προσλήψεις που χρειάζονται και πώς θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και τα νέα εργαλεία που θα τους δοθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάθε νομοθέτη. Όλα αυτά πρέπει να τα ακολουθεί. Όταν θεσπίζουμε νομοθεσία, που είναι δύσκολο αυτό, θα πρέπει να φροντίζουμε και να εφαρμόζεται την νομοθεσία αυτή. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα εδώ πρόκειται για θέμα ομοφωνίας με το Συμβούλιο. Αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολλή δουλειά να κάνει. Βλέπετε τη δουλειά που γίνεται στις ε, επιτροπές και εδώ και πρέπει να γίνει και ένα follow-up, μια παρακολούθηση της υπόθεσης για να εξασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία θα εφαρμόζεται υπέρ των ε, φορολογουμένων που πληρώνουν τους φόρους. Ο Μπέρναρ Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την τελευταία σας απάντηση, γιατί ε, από την εμπειρία μας, από την ε, Επιτροπή Πανά και την τάξη 1 και 2, βλέπουμε ότι τα κράτη είναι ε, απρόθυμα να ασχοληθούν με τις επιμέρους περιπτώσεις. Αναφέρατε παραδείγματα αλλαγών. Θα σας παρακαλούσα ή θα πρότεινα, πέρα από τις επιμέρους υποθέσεις που υπάρχουν πάρα πολλέ στα Panama Papers, Paradise Papers. Πέρα από αυτά να ε, δείτε και το θέμα του blacklist του κυρίου Μορφσκοβισή και να υποβάλλετε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όχι μόνο να λύσετε εκ των υστέρων περιπτώσεις ε, για το πώς μπορούν να αλλάξουν οι ε, αθέμητοι όροι ε, του ανταγωνισμού. Τώρα, οι ε, εκ των προτέρων άδειες ε, για επιδοτήσεις. Θέλω να αναφερθώ σε έναν Κινέζο επενδυτή σε αεροδρόμιο. 100 εκατομμύρια ε, επιδοτήσεις δόθηκαν για το μέλλον, μέχρι το 2024. Πάνω στη βάση ενός άγνωστου επιχειρηματικού μοντέλου και πάνω στη βάση δεδομένων ε, από τον πολιτή για δημιουργία θέσεων εργασίας που δεν ελήφθη. Ανέφερε ότι θα ήταν εξασφαλισμένες 11.000 θέσεις εργασίας, ενώ στην πραγματικότητα ήταν 2.000. Ε, τι εξέταση γίνεται προκειμένου να δοθούν εκ των προτέρων άδειε. Μιλήσατε για τη Lufthansa Air Berlin. Αν ισχύει η 4η Δεκεμβρίου και αν αυτή είναι η ημερομηνία, εντάξει. Αυτή τη στιγμή 120 αεροπλάνα της Air Berlin δεν πετούν, περιμένοντας την απόφαση της Κομισιόν, από ό,τι λένε, και εγώ ε, είδα και από τη Φραγκφούρτη για το ε, Βερολίνο ε, πετούν αεροπλάνα 747. Η ε, παρατήρηση για τη Ryanair δεν ισχύει. Οι πιλότοι δεν έχουν ε, σωστές συμβάσεις, ε, είναι τελείως άδικες οι συνθήκες εργασίας και φεύγουν από εκεί. επίσης, στη Ρινανία Παλατινάτο, στη τράπεζα ε, αποκάλυψε ότι δημιουργήθηκαν ε, ψεύτικες εικονικές επιχειρήσεις ε, που δραστηριοποιήθηκαν σε συνταξιδοτικά προγράμματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και θα πρέπει να γίνει έλεγχος των κανόνων ανταγωνισμού. Από πού να το πιάσω. Για το τελευταίο, το παρακολουθούμε αλλά δεν έχω τίποτε καινούριο. Θα επανέλθουμε όμως. Για τη φερολογία και να το κλείσω αυτό το θέμα. Προσπαθούμε ακόμα και αυτή είναι η δουλειά μας να δώσουμε καλύτερη καθοδήγηση γιατί είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις που εξετάζουμε, αλλά και γενικότερα λέμε να αυτή είναι η προσέγγιση με την καθοδήγηση. Και καμιά φορά μας λένε κάποιοι, α, είναι καινούριο όλα αυτά, νέες, νέες ε, ερμηνείες κτλ. Όχι. Και το δικαστήριο δίνει καθοδήγηση. Το 1998 δεν είχε δώσει που έλεγε ότι μπορεί να έχει κρατική ενίσχυση, διαφορές μορφές, φορολογικές κτλ. Ένα αυτό. Δύο, μπορεί να υπάρχουν συναλλαγές εντός ενός ομίλου, αλλά αν θέλει κανείς να είναι και ε, ασφαλή σε σχέση με τον ανταγωνισμό, πρέπει να δίνει τιμές αγοράς και για τις ενδοομιλιακές συναλλαγές. Υπάρχουν λοιπόν οι βασικές οδηγίες, οι αρχές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις, ε, η φοροτεχνική και ούτω καθεξής. Και το λέω αυτό με απόλυτη ασφάλεια γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν γίνει φορολογικές ρυθμίσεις τύπου tax rulings που ήταν σύμφωνες με τον ανταγωνισμό γιατί τα κράτη ξέραν τι κάνανε και δεν, έκαναν, δεν παραβιάζαν τον ανταγωνισμό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να εξετάσουμε και δεν υπάρχει καμιά ανησυχία ή μέλημα διότι κάνουν καλή δουλειά τα κράτη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ισχύει πάντα. Για τα αεροδρόμια. Στην περίπτωση των μεγάλων αεροδρομίων υπάρχει το λεγόμενο plain vanilla path που έχει να κάνει με το σχεδιασμό και την πιστοποίηση. Αλλά υπάρχουν και τα μικρότερα αεροδρόμια που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τον κανονισμό γενικής εξαίρεσης ε, αποκλεισμού ώστε να μην υπάρχει μία απόφαση εδώ και 50 εκεί. Εμείς μπορούμε έτσι να παρακολουθούμε καλύτερα που είναι τα μελήματα τα σχετικά με τον ανταγωνισμό ή τα προβλήματα τους. Λέμε δηλαδή να υπάρχει μια γενική συνταγή για τις κρατικές ενισχύσεις. Εάν το κάνετε αυτό όπως σας το λέμε, δεν χρειάζεται να το κοινοποιήσετε στην Επιτροπή. Βέβαια, αποφάσεις που λαμβάνονται υπό το Γενικό Κανονισμό Εξαίρεσης Αποκλεισμού. Κάνουμε και ένα δημοτολογικό έλεγχο για να βεβαιωθούμε ότι όλα πάνε καλά. Αλλά ο κανονισμός έχει λόγο ύπαρξης το να δώσει μια αυτόνομη δυνατότητα δράση στα κράτη-μέλη. Και να λένε ναι, κάνουμε αυτή και αυτή την επιλογή, μπορεί να έχουμε αυτό και αυτό το πρόβλημα τα κράτη, αλλά με την Επιτροπή δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε στις ρυθμίσεις μας χωρίς να ανησυχούμε τι θα μας πει η Επιτροπή. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση του Κινέζου επενδυτή δεν έχω να σας πω. Κάτι δεν τη γνωρίζω. Αλλά σε παρένθεση θα επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει νέα εργαλεία για ε, διερεύνηση, επισκόπηση των επενδύσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή λύση και για τις ε, ξένες άμεσες επενδύσεις. Μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε λοιπόν καλύτερα εργαλεία από εδώ και μπρος και με αυτό το εργαλείο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφτηκα την Κίνα για να συζητήσουμε πώς θα δώσουμε νέα ουσία ε, στον ε, τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το διαρθρωμένο διάλογο για τις ε, επενδύσεις. Να είναι πιο απλά και ξεκάθαρα τα πράγματα. Τι εννοούμε όταν λέμε θεμητός ανταγωνισμός. Και εν τέλει για την Air Berlin. Ο λόγος για τον οποίο άλλαξε η αγορά ήταν ότι πτώχευσε η Ερπελίν. Δεν έφταιγαν οι έρευνες της Επιτροπής. Η εκκρεμότητα μιας απόφασης από την Επιτροπή ήταν η πτώχευση της Ερπελίν. Αυτό κατέβαζε το αεροπλάνο στο έδαφος και τα κράτησε στο έδαφος. Και ε, η συνέπεια που βλέπουμε είναι αλλαγές στις τιμές που αποφασίζουν οι εταιρείε των οποίων τα αεροπλάνα εξακολουθούν να πετάνε. Επομένω, η εξαίρεση για τα αεροπλάνα που είναι καταχωρημένα και μάλιστα πλήρη, με, με πλήρωμα δηλαδή, wet listed, ε, αυτό το νόημα έχει να, να μείνουν στον αέρα τα αεροπλάνα με την Air Berlin πριν, με την Lufthansa τώρα, να μπορούν να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, ε, ο πελάτης να μην βρεθεί ε, να έχει χάσει το, το ειστήριό του ή να μην έχει την εξυπηρέτηση στο δρομολόγιο του. Ευχαριστώ Περβάνος Περές. Σας ευχαριστώ. Πολλά θέματα τέθηκαν. Αλλά δεν είπατε τίποτα για τη McDonald's ακόμα. Τι γίνεται με την έρευνα για τα McDonald's. Λένε επίσης ότι οι υπηρεσίες σας έχουν κάνει ερευνητικές επιτόπου προσπάθειες για να δουν με ποιο τρόπο έδιναν την δυνατότητα για κάποιες ενέργειες euh, πώς ε, τήρουσαν τα fintech από πλευρά ορισμένων τραπεζών και επίσης τι γίνεται και με τον ρόλο που μπορεί να παίξουν οι κρατικές επιδοτήσεις στον τομέα του διεθνούς ανταγωνισμού. Το καθεστώς ε, ε, αυτό είτε στα πλαίσια του ΟΣΑ είτε στα πλαίσια του ΠΟΕ είναι κάτι το οποίο δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση ε, των προβλημάτων αυτών και της χρήσης των επιδοτήσεων των κρατικών ανάμεσα στις διάφορες χώρες και στο εσωτερικό της Ένωσης και στο εξωτερικό της Ένωσης. Οι απαντήσεις φυσικά θα πρέπει να αναζητηθούν και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί από αυτά τα θέματα θα εξαρτηθεί η μελλοντική σχεδίαση της πολιτικής ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας δεν το κατάλαβα, λέει η κυρία Βέσταγκερ. Όχι το Μακδόναλντ, όχι το τελευταίο κομμάτι. Λέω για σε σχέση με το FinTech, τις έρευνες που κάνατε στα πιστοτικά ιδρύματα, τίποτα άλλο. Δεν έπρεπε να ρωτήσω. Δεν έπρεπε να Δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σας γιατί μετά θα σταματήσει η διευμηνία. Κοιτάξτε, δεν έχω ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα. Θα επανέλθουμε κάποια άλλη φορά. Διερευνούμε πάντως ακόμα και τώρα τα McDonald's. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση αυτή. Εξ αρχής είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι νομίζαμε στην αρχή. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις σχέσεις ε, με τις ε, συμφωνίες αποφυγής ε, διπλής φορολογίας. Θα πρέπει να βεβαιώσουμε την νομική μας εδώ θέση. Θα επανέλθουμε όμως το ταχύτερο δυνατόν. Για την τελευταία ερώτηση σε σχέση με τις κρατικές επιδοτήσεις αυτό είναι ένα κομμάτι θα έλεγα της ε, διεθνούς μας στρατηγικής το οποίο ε, θεωρώ ότι είναι κρίσιμο. Ήμουνα στην Κίνα την προηγούμενη εβδομάδα και το λέω αυτό γιατί στις κινέζικες αγορές αποφάσισαν να εφαρμόσουν έναν μηχανισμό ελέγχου του υγιούς ανταγωνισμού. Εφαρμόζεται τον τελευταίο χρόνο και σε κρατικό επίπεδο, συγκεντρωτικά δηλαδή, και σε επίπεδο περιφερειών. Στην ουσία εξετάζουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις για να δούνε σε ποιο βαθμό η πολιτική του ανταγωνισμού γίνεται σεβαστή στις αγορές. Για μας αυτό ήταν ένα σημείο εκκίνησης για ένα μνημόνιο κατανόησης έτσι ώστε να συζητήσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο τις κρατικές επιδοτήσεις. Ε, τώρα προσπαθούμε να δούμε σε ποιους τομείς θα γίνουν οι πρώτες έρευνες. Ε, έχουμε συζητήσει ε, πολύ το θέμα του χρηματοπιστωτικού τομέα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Κίνα γύρω από αυτό τον τομέα και ίσως να έχουμε και εμείς κάτι να προτείνουμε. Έχουμε φτάσει τα 700 στα τα τελευταία 10 χρόνια στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Δηλαδή και εμείς δεν είμαστε άγιοι σε σχέση με τις κρατικές επιδοτήσεις. Εάν λοιπόν είμαστε επιτυχείς στη συνεργασία και με τις υπόλοιπες πλευρές εκτός Ένωσης, θα βρούμε, θα έλεγα, περισσότερα επίπεδα διαφάνειας που θα μας ικανοποιήσουν. Δεν γίνονται αυτά δια Αυτό θα γίνει και στα πλαίσια του ΠΟΕ, ε, είχαμε αρκετά σημεία επιτυχίας αν θέλετε στις προσπάθειες μας στο ΠΟΕ αλλά καθυστερούμε πάρα πολύ. Σαν παράδειγμα στις αγροτικές εξαγωγές ε, είχαν συζητήσει εδώ και δύο χρόνια ε, και είχαν πάρει κάποιες πρώτες αποφάσεις. Η συζήτηση όμως είχε ξεκινήσει πριν 15 χρόνια. Το θέμα είναι λοιπόν να βρούμε τρόπο έτσι ώστε όταν συνάπτουμε διμερείς εμπορικές συμφωνίες να ξέρουμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά και στην εμπορική συμφωνία με την Νότια Κορέα και στην εμπορική συμφωνία με τον Καναδά. Θα πρέπει να σπάσουμε το ταμπού των κρατικών επιδοτήσεων. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί γιατί βλέπουμε ότι οι ορισμένους τομείς είναι θεμητοί η κρατική επιδότηση. Σε άλλους τομείς αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισμού. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να δίνουμε χρήματα στην εκπαίδευση, στην καινοτομία, στα κοινωνικά θέματα, στην εκπαίδευση. Ε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και αυτό θα μας βοηθήσει θα έλεγα στο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά στο μέλλον. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πάντως ξεκίνησε και ξεκίνησε με διαρθρωτικό και συγκεκριμένο τρόπο. Και έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε Σχετικά με τις προμήθειες, σαν παράδειγμα, ε, παίζουν ρόλο όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Ε, και θα πρέπει ε, γενικότερα όλα τα θέματα που άπτονται ε, της πολιτικής ε, των επιδοτήσεων των κρατικών να τεθούν υπό συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ Επίτροπε, λέει ο κ. Γκουαλτιέρη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων μαζί σας η συνεργασία μαζί σας θα συναχιστεί. Θέλω να ευχαριστήσω και την διερμηνία. Κλείνουμε την Πέμπτη έχουμε μία συνάντηση στις 8.30 το πρωί μαζί με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και στις 9 και 4 την τακτική μας συνεδρίαση.